Αγαπητοί συνάδελφοι, α ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Έχουμε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να το εγκρίνουμε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 22ης και 23ης Μαρτίου 2017 μπορούν και αυτά να εγκριθούν αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει και δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση μας αυτή με την ε, Επίτροπο κυρία Μπούλτσα, την οποία έχουμε την τιμή να έχουμε ανάμεσά μας, για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018. Χαίρομαι όλους ιδιαιτέρως, κύριε Επίτροπε, που είστε δίπλα μου, διότι ε, συνεργαζόμαστε πολύ συχνά και πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά να σε έχουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, διότι ξέρετε ότι ήδη έχουμε συνεργαστεί στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου, οπότε βρισκόμαστε και σε συνεχή επαφή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά φέτος έρχεστε να μας δείτε εδώ, στην Επιτροπή Μεταφορών. Στόχος του διαρθρωμένου αυτού διαλόγου είναι να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, και στόχος είναι να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργασία μας για το 2018. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, κυρία Επίτροπε, θα σας ήμασταν ιδιαίτερα ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας διαφωτίσετε ήδη από τώρα για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018, στο πλαίσιο βέβαια της πολιτικής μεταφορών. Στόχος λοιπόν της σημερινής συζήτησης να καταφέρουμε να λύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα που έχουμε από την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 Ξέρετε ότι πολύ συχνά ταινίζουμε μόνο το μέλλον, αλλά ξεχνάμε λίγο ότι έχουμε και κάποια σημαντικά επιτεύγματα πετύχει. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να τα θυμόμαστε αυτά, να κάνουμε έναν απολογισμό. Προφανώς παραμένει ακόμα να γίνει πολλή δουλειά προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο πλαίσιο τη πολιτική μεταφορών. Και βέβαια γνωρίζετε όλοι, ότι όλοι στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής θέλουμε ασφαλείς, αποτελεσματικές και προσιτές μεταφορές, οι οποίες θα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση στα πλαίσια της ψηφιακής ανάπτυξης, να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη παγκόσμια συνδετικότητα. Τίθεται βέβαια παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα, θα πρέπει να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ή να δημιουργήσουμε και νέε θέσει απασχόληση και τίθεται βέβαια και το ζήτημα του περιβάλλοντο και τη προστασία του περιβάλλοντο. Μιλάμε όλο και περισσότερο για τι κλιματικέ αλλαγέ και τι σχετικέ προτεραιότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν το περιβάλλον. Κύριε Επίτροπε, θα σα δώσω το λόγο τώρα για 10 λεπτά, θα μα κάνετε μια παρουσίαση. Στη συνέχεια είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε μια πολύ δυναμική επικοδομητική συζήτηση με τα μέλη τη Επιτροπή μα και θα αλλάξουμε τώρα και λίγο τη μέθοδο μας, κύριε Επίτροπε. Δηλαδή, μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου, θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές για πέντε λεπτά, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση λεγόμενη ping-pong. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πιο δυναμική συζήτηση. Θα είναι πέντε όμως μόνο τα λεπτά τα οποία θα έχετε. Αυτό θα είναι το ανώτατο όριο. Πέντε λεπτά δηλαδή τα οποία μπορείτε να επιμεριστείτε με την Επίτροπο προκειμένου να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να τεθούν ερωτήσεις και να ακουστούν απαντήσεις και ενδεχομένω να θέσετε και νέες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρουν και άλλα μέλη της Επιτροπής μας για τρία λεπτά αυτή τη φορά ο καθένας. Κυρία Μπούλτσα, Πρέπει να σας πω ότι το να έχουμε δύο γυναίκες στα δύο αυτά θεσμικά όργανα και να λέμε ότι εργαζόμαστε πολύ επικοδομητικά και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση για ζητήματα τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για μας, με τέτοια ενέργεια, με τέτοιο ενθουσιασμό, θα έλεγα πραγματικά είναι πραγματική περηφάνεια αυτό για μένα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα στην Επιτροπή μας και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Καρίμα, αγαπητή Αντιπρόεδρε, εξότιμα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, κυρίες και κύριοι, έχουμε και προσκεκλημένους από ό,τι βλέπω, τους καλωσορίζω και αυτούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά. Ουσιαστικά η παρουσίασή μου θα αποτελείται από δύο κύρια τμήματα. Το πρώτο η επισκόπηση της υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και το δεύτερο τμήμα είναι να δούμε προς το μέλλον. Θα σας παρουσιάσω επομένως ε, το πρόγραμμα εργασίας ε, που αρχίζουμε να σχεδιάζουμε για το 2018 και αν μου επιτρέπετε περνώ ευθύ αμέσω στο συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα το πακέτο κινητικότητας είναι ο σημαντικότερος στόχος μας ε, να παραδώσουμε τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα το 2017 και θα έχουμε τη δυνατότητα το θέμα να το συζητήσουμε και στην προσεχή Σύνοδο Ολομέλειας, όπου και θα παραστώ για να, μάλλον και θα παραστώ στην Επιτροπή σας 19 Ιουνίου για να σας παρουσιάσω ακριβώς ε, τις λεπτομέρειες των προτάσεων της Κομισιόν. Σήμερα μια σύντομη ενημέρωση για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξεκίνησε ως μικρότερο πακέτο, ε, το οδικό πακέτο όπως λεγόταν, πλέον έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει εγκάρσια στοιχεία. Ε, προσπάθεια της Κομισιόν είναι να καταπολεμήσει τα στεγανά. Και στις μεταφορές θέλουμε ε, να έχουμε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα. Το πακέτο κινητικότητας θα περιλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες για τον, οδικό, για τον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά και προτάσεις όπως παραδείγματος χάρη πρότυπα για τις εκπομπές του άνθρακα για τα φορτηγά οι πρώτε 7 προτάσει θα είναι έτοιμε για έγκριση σε 4 εβδομάδε, την 31η Μαου, ενώ θα ακολουθεί στα τέλη του έτου περίπου μια δεύτερη δέσμη προτάσεων. Πιστεύω ότι θα θεωρήσετε κι εσεί ε, ότι είναι άρτιο και ισορροπημένο αυτό το πακέτο κινητικότητα ε, με έντονε κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ, ψηφιακέ πτυχέ, πτυχέ που άπτονται τη εσωτερική αγορά, ε, με στόχο τη μείωση τη γραφειοκρατία, η βασική μα προτεραιότητα άλλωστε, και δεύτερον ενισχύουν την επιβολή, την εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το σχέδιο ψηφίσματο για το θέμα αυτό που είχατε εγκρίνει στην Επιτροπή σα πριν από ορισμένε εβδομάδε. Όμω εδώ χρειάζομαι τη δική σα βοήθεια και σα παρακαλώ να ασκήσετε πίεση στα κράτη-μέλη, τα οποία και αυτά πρέπει να προσχωρήσουν στι προσπάθειέ μα ε, και με ανοιχτό τρόπο ε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και βέβαια να τα εφαρμόσουμε όπω ε, έχουμε συμφωνήσει. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι προτάσεις αυτές έχουν μεγάλη πολιτική σπουδαιότητα και θα είναι σημαντικό να συνεργαστούμε ώστε πραγματικά το πακέτο στο σύνολό του να μπορέσει να γίνει δεκτό ε, στη διάρκεια της θητείας μου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα εξασφαλίζει και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Βασίζομαι σε εσά λοιπόν για να αντιμετωπίσετε τις προτάσεις αυτές ως προτεραιότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να ορίσετε και τις δικές σας ομάδες εγκαίρως ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εντός ε, των ε, πλησίων και προθεσμιών που προβλέπουμε. Δεύτερο θέμα, δική ασφάλεια. Αλλά πρώτα, αφού είμαστε, γιατί, επειδή είμαστε λοιπόν σε οδικές μεταφορές, να μιλήσω για την οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα που παρουσίασα στην ε, Βαλέτα ήταν και πρόεδρος ε, παρούσα και ορισμένοι από εσά. Ο στόχος ήταν ε, να, μειώσουμε ακόμη περισσότερο του θανάτους από τροχέα. Είχαμε 2% μείωση στα μοιραία στα αλλά 25.000 500 ε, άνθρωποι, παρότι είναι πολύ δύσκολο να μιλά κανείς για νούμερα για αυτά τα θέματα, χάνουν τη ζωή τους. Έχασαν τη ζωή του το 2016. Συγκεκριμένα 600 λιγότεροι από το 2015, 6.000 λιγότεροι από το 2010 ενθαρρυντική διαφορά αυτή από το 10 στο 16, 6.000 λιγότεροι θάνατοι. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό, εφόσον έχουμε επίσης και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών, σοβαρών τραυματιών, 135.000 άτομα το χρόνο, με βάση τα τελευταία στοιχεία. Την 1η Φεβρουαρίου λοιπόν εγκρίναμε μια πρόταση για τροποποίηση τη οδηγία ε, που θεσπίζει τι απαιτήσει εκπαίδευση για του επαγγελματίε οδηγού που θα συνεισφέρει σε πιο υψηλά πρότυπα οδική ασφάλισης στου επαγγελματίε οδηγού. Ε, Μα κινητοποίησε το ότι το 10% ε, είναι από φορτηγά ε, και το 10% από τα βαν. Και πρέπει να τα αποκριθούμε. Το Συμβούλιο ήδη έχει εξετάσει την πρόταση σε πρώτη ανάγνωση. Ήταν πολύ επικοδομητική η προσέγγιση και το καλωσορίζω αυτό. Περιμένουμε λοιπόν να συνεργαστούμε και το δικό σα συζητητή, τον κύριο Λούντγκρεν, του Σκιώδη και το Κοινοβούλιο εν γέννη, ώστε να εγκριθεί το σημαντικό αυτό νομοθέτημα. Είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή σα θα δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο θέμα τη οδική ασφάλεια. Το επόμενο θέμα είναι η αεροπορία. Για το 2017 πάντα. Περνάμε λοιπόν στον τομέα της αεροπορίας. Εδώ προετοιμάζουμε ε, μία δέσμα θετικών μέτρων για την ε, αέρια συνδεσιμότητα που θα απογειωθεί νωρίς, όπου να είναι, σε 7 Ιουνίου. Και με αυτή τη δέσμη μέτρων εφαρμόζουμε ε, τη στρατηγική για την αεροπορία, περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τι υποχρεώσει δημόσια υπηρεσία, ιδιοκτησία, έλεγχο και περιλαμβάνει και μια νομοθετική πρόταση για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού στι ενέργειε μεταφορέ, αντικαθιστάται τον κανονισμό 868 2004. Είναι μια νομοθετική πρόταση που έρχεται ε, κατόπιν δικού σα αιτήματο, ε, ε, του Κοινοβουλίου δηλαδή που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στη διάθεσή της ένα αποτελεσματικό εργαλείο δράσης για την αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών τρίτων χωρών σε βάρος των αεροπορικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη ε, έχουν σας απόψεις μεταξύ τους και εδώ ζητώ πάλι τη δική σας υποστήριξη να έχετε κι εσείς εδώ μια τις συζήτηση στο επίπεδο της Επιτροπής σας αλλά να μπορέσετε να ασκήσετε πυρού και στο εθνικό επίπεδο. Έρχομαι τώρα στην ε, ΕΑΣΑ, ε, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Αεροπορία. Ο νέος κανονισμός είναι μια ευκαιρία να κάνουμε το σύστημα της ενέργειας ασφάλειας πιο αποτελεσματικό. Κάντε κι εσείς λοιπόν μια ακόμη προσπάθεια για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν το νομοθέτημα αυτό. Γιατί μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό τη Ευρωπαϊκή Αεροπορία. Παρακαλώ να εστιάσετε την προσοχή σα όσο το δυνατόν περισσότερο και σε αυτό το σημείο. Το 2017 πάντα για τα σιδηροδρομικά. Εδώ προτεραιότητα για φέτος και του χρόνου είναι η υλοποίηση της φυστάμενης νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες μου βάζουν τις τροχές τώρα για να επεξεργαστούμε την ενίσχυση, την, ε, συγγνώμη, την εφαρμογή της αναδιατυπωθήσης οδηγίας και το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους ώστε να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για το άνοιγμα της αγοράς το 2019. Παραδείγματο χάρη θέλουμε εκτελεστικές πράξεις ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ε, εγκαταστάσεις δρομικών υπηρεσιών όλοι οι φορείς μετάλλευσης, ε, σταθμοί επιβατών, παραδείγματο χάρη και επίσης θέλουμε να εξασφαλιστεί η οικονομική ισορροπία των συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών. Θέματα που ξέρω ότι ενδιαφέρουν πολύ την δική σας Επιτροπή. Να πω δύο λόγια για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει την πρότασή της για το θέμα αυτό πριν από το καλοκαίρι. Εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα στον ε, ισχύοντα κανονισμό Δηλαδή είχαμε κάποιες εμβαλωματικές εφαρμογές, παρεκκλήσεις, ε, δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου. Γι' αυτό και θέλουμε να διευκρινίσουμε ε, ακόμη περισσότερο τους υφιστάμενους κανόνες. Στόχος μας είναι να ορίσουμε καλύτερα την έννοια της έκδοσης εισιτηρίων μέχρι τον τελικό προορισμό, through ticketing και, και τις ε, σχετικές υποχρεώσεις για τις συνδρομικές επιχειρήσεις και τους πολιτές εισιτηρίων. Θέλουμε επίσης να προτείνουμε την εισαγωγή μιας ρήτρας ανωτέρας βία. Ε, για να συμμορφούνται και προς τις άλλες, ε, άλλα νομοθετήματα. Επίσης το 2017 είναι το έτος ε, της θάλασσας και της ναυτιλίας. Έχουμε διαβουλεύσεις με τους, όλους τους ενδιαφερομένους για τις προτεραιότητες, για τον τομέα, για να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και ποια είναι η απαραίτητη εξέλιξη στο θέμα των πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε νέε νομοθετικέ πρωτοβουλίε το 2018, αν συμφωνείτε. Μπορώ να πω και λίγο περισσότερα πράγματα. Ήδη φέτο όμω έχουμε την αναθεώρηση τη οδηγία για τι εγκαταστάσει ε, υποδοχή των λιμένων. Θα συνεχίσουμε επίσης το έργο μας για την ε, πανεξέταση τη νομοθεσία για τι θαλάσσιες μεταφορέ. Η στόχη μα είναι ξεκάθαρη. Ξεολόγηση του κανονισμού για την ευθύνη ε, των ε, μεταφορέων επιβατών στη θάλασσα περίπτωση ατυχήματος, αξιολόγηση του REFIT σε σχέση με την νομοθεσία για την εκπαίδευση και επιστοποίηση των αυτών και επίσης το ναυτικό check-up που θα καλύπτει τις ευθύνες του κράτους σημαίας, ε, τον έλεγχο του κράτους λιμένος και τις απαιτήσει για το παράκτιο κράτος. Πολύ σύντομα τώρα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πολύ καλή πρόοδο που έχετε σημειώσει όσον αφορά τα αρχή ασφάλειας επιβατηγών πλοίων και όσον αφορά τις εκθέσεις τις οποίες εγκρίνατε τον Απρίλιο αφού καταφέρατε να καταλήξετε σε συμβασμούς για κάποια πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων τριμερών διαλόγων. Τώρα το επόμενο θέμα μας είναι η απαλλαγή από τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε ότι οι μεταφορές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν για να αντιστοιχούν περισσότερο στη ζήτηση, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο βιώσιμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενεργειακά αποδοτικές, απαλλαγμένες από τις ανθρακούχες εκπομπές μεταφορές. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και προβλέπει για φέτος νέα μέτρα. Η οδηγία για τα αναλλακτικά κάψιμα θα δέωσε εμπιστοσύνη στην βιομηχανία, του επενδυτέ και του καταναλωτέ και καλό όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων πολιτική. Στο τέλο του έτου, ω δεύτερο τμήμα τη νομοθετική δέσμη για την κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σκεγγραφίσει τα μέσα υποστήριξη για ένταξη στην αγορά οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών λεωφορείων θα προβλέπεται επίση αναθεώρηση τη οδηγία για τι δημόσιε προμήθειε καθαρών οχημάτων και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελέσει η οδηγία αυτή μια κινητήρια δύναμη για καινοτόμα προϊόντα. Τέλο, θα έχουμε και μια πρόταση για συνδυασμένε μεταφορέ, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια αλλαγή του τρόπου εκτέλεση των μεταφορών από τι οδικέ εμπορευματικέ μεταφορέ προ τι θαλάσσιε μεταφορέ μικρών αποστάσεων ή τι αεροδρομικέ μεταφορέ. Θα ήθελα να πω κάτι για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορώ, κυρία Πρόεδρε, γιατί από ό,τι φαίνεται εξάτλησα το χρόνο που μου είχατε δώσει. Είναι πολύ σημαντική η χρηματοδότηση μεταφορέ. Πρέπει να έχουμε επενδύσει λοιπόν σε υποδομέ και αυτό αποτέλεσε προτεραιότητα του Πρόεδρου Γιούγκερ. Ενώ προβλέπεται ότι προβλεπόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτίμαζε μία πρόταση για το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι τα τέλη του 2017, από ό,τι φαίνεται τώρα μία λεπτομερή πρόταση θα ολοκληρωθεί μόνο στι αρχέ του 2018. Το νέο σημαντικό όμω ορόσημο είναι η συζήτηση προσανατολισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2025. Εν συνεχεία, Τη της Λευκής Βίβλου συζήτηση που θα ξεκινήσει 28 Ιουνίου 2017. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και να προωθήσουμε την εξαιρετική πορεία που είχε ακολουθήσει ο μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Την περίοδο 2016-2016, 37,6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικών επενδύσεων κινητοποιήθηκαν με 20 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων που συνέβαλαν στο θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Προσβλέπουμε σε μια συνεχιζόμενη υποστήριξη προ την κατεύθυνση αυτή. Προβλέπεται όμω ότι 740 δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται ακόμα προκειμένου να έχουμε ένα κεντρικό δίκτυο των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και προκειμένου να απαλληφθούν οι κύριοι παράγοντε συμφόρηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε κινητοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το επενδυτικό μοντέλο για την Ευρώπη και σήμερα βλέπουμε ότι οι 36 δράσεις που κινητοποίησαν συνολικά 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχετικές επενδύσεις έχουν ήδη επιτευχθεί. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά μας ενθαρρύνει για τη μελλοντική μας εργασία. Τέλος, προβλέπεται μια νέα πρόταση υποβολής προσφορών για συνδυασμένη χρηματοδότηση στο σκέλος μεταφορών του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη και κατά αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε καλύτερη μόχλευση. Τώρα, το πρόγραμμα εργασία για το 2018, πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτροπικότητα. Το 2018 θα είναι πραγματικά το έτος της πολυτροπικότητας. Θα βελτιώσουμε την ενσωμάτωση όλων των μέσων μεταφοράς στο γενικότερο δίκτυο μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά νέων προτάσεων για τι θαλάσσιε μεταφορέ που θα προκύψουν από τον έλεγχο καταλληλότητα, το fitness check για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Όσον αφορά τι θαλάσσιε μεταφορέ, το πιο σημαντικό ζήτημα θα είναι η αναθεώρηση των διατυπώσεων υποβολή δηλώσεων. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε εδώ πέρα στα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει μια ενιαία ευρωπαϊκή θηρίδα, συμπληρωματική ω προ τι εθνικέ ενιαίε θηρίδε άλλα ζητήματα μας απασχολήσουν θα είναι ο έλεγχο του κράτους σημαίας και του κράτους λιμένε, παρακολούθηση της κίνησης των πλοίων, καθώς επίσης και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των ναυτικών. Όλα αυτά αποτελούν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας νομοθεσία του Πρόεδρου Γιούγκερ. Θέλουμε επίσης να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε, να μειώσουμε μάλλον τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ήδη από τον Άνοιξη του 2018 να έχουμε συγκεκριμένου στόχους μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μετά την διάσκεψη για την οδική ασφάλεια στη Μάλτα το Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής όσον αφορά την οδική ασφάλεια για όλο το χρονικό διάστημα μετά το 2020. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίνανε το 2017, αυτά τα οποία προβλέπουμε ότι θα γίνουν το 2018, και ελπίζω ότι θα έχω και τη δική σας υποστήριξη για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και προσβλέπω βέβαια σε περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία μαζί σας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, οπότε κυρίως από την άρεξη της συζήτησης. Στη μέθοδο την καταλάβατε, έτσι. Έχετε ο καθένας πέντε λεπτά μετά τα πέντε λεπτά κλείνω το μικρόφωνο, έτσι σας έχω προειδοποιήσει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πεντάλεπτο έχετε τη δυνατότητα να έχετε την απάντηση τη Επιτρόπου. Άρα, όσο πιο σύντομες ερωτήσει κάνετε, τόσο περισσότερο χρόνο θα αφήσετε για την απάντηση στην Επιτρόπου. Ο κύριο Βιμ Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή ε, το ότι ξεκινάει με μένα η νέα αυτή η συζήτηση με ερωτοποκρίσεις και η πρώτη ερώτηση είναι θα έρθει εγκαίρο το πακέτο κινητικότητα. Πρέπει να σα πω ότι το περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό και είναι πολύ ε, γοητευτικό το ότι ζητάει τώρα γρήγορη δουλειά η Επίτροπος από το Κοινοβούλιο, αλλά το ερώτημα είναι εάν θα έρθει εγκαίρος. Ε, υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις αντικτύπου, εάν κατάλαβα καλά. Πρέπει να δούμε και το better regulation του κυρίου Τίμερμανς. Πρώτη ερώτηση. Θα έρθει εγκαίρως. Πρώτα απ' όλα, ελπίζω να αναγνωρίσουμε από κοινού ότι δεν χάθηκε ο χρόνος γιατί υπάρχει και ένας νέος τρόπος προετοιμασίας των νομοθετικών προτάσεων, δηλαδή με διαβούλευση για να μιλήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν ε, ξεκινήσει η διαδικασία. Οπότε για να σας ε, τα πω λίγο θεωρώ ότι μπορούμε, είμαστε εντός ε, του προγράμματος που έχουμε θέσει και μπορώ να σας αναφέρω και κάποια σημεία που θα ενισχύσουν την άποψη. Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, διαβουλεύσει όλους τους ενδιαφερόμενους και κοιτάμε ακριβώς τον πιθανό αντίκτυπο των μέτρων και η Προεδρία, Εστονία, Βουλγαρία και Αυστρία είπαν ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν στο πακέτο κινητικότητας και θα αποφασίσει ο καθένας ποιο κομμάτι του πακέτου κινητικότητας θα αποφασιστεί από ποια Προεδρία. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να αποτελεί περαιτέρω εγγύηση και ελπίζω ε, ότι μπορώ να βασιστώ και πάνω σας. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο στοιχείο. Η Κομισιόν ε, έκανε αυτό που πρέπει, το Συμβούλιο λέει ότι θα το κάνει και ελπίζω να ακούσω και μια ανάλογη δέσμευση από σας. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή για την κοινωνική παράγραφο. Είναι παντού στις εφημερίδες έχουν διαρρεύσει κάποια σχέδια, ανησυχούν τα συνδικάτα. Έχουμε συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης που είναι πραγματικά πολύ ανήσυχοι. Μιλήσατε εσείς με τα συνδικάτα. Τι τρέχει με τα κοινωνικά ζητήματα. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει αυτή η ανησυχία στις εφημερίδες παντού. Και υπάρχει αμφιβολία τελικά για το πακέτο. Δυστυχώ πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας, λέει ο Επίτροπο. Και ο λόγος για τον οποίο μου προξενεί έκπληξη είναι το ότι η δικιά μα πόρτα είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να μας μιλήσει για να δούμε αυτό το ζήτημα, ειδικά την κοινωνική πτυχή και ανησυχώ για το ότι διάφοροι διασπείρουν φήμες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα όσα υπάρχουν στο πακέτο όταν άκουσα για πρώτη φορά και είδα δηλαδή κάτι βολάν που μοίραζαν τα συνδικάτα, πήγα να τους δω όταν ε, συναντήθηκαν δίπλα στον Περλεμόν. Και τους μίλησα και τους μίλησα το απόγευμα και ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή από τα έξι πράγματα που λέγανε, τα έξι τα έχουμε ήδη δει στο πακέτο, όπως ε, θέλανε. Το ένα ακόμα είναι υποδιαπραγμάτευση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σφόρουμε 100% στα πάντα. Αλλά υποσχέθηκα στον κύριο Ερτούγ ε, στο πρώτο έτος εντολής ότι θα περιληφθούν τα κοινωνικά ζητήματα, ότι θα τα δούμε συστηματικά μαζί με τα άλλα θέματα. Ε, πραγματικά θα ήθελα να σας προσκαλέσω και εσάς. Ε, μην διασπείρετε φήμες. Φήμες οι οποίες βασίστηκαν στην ε, δημόσια διαβούλευση, όπου βεβαίως ε, ε, μαζέψαμε όλες τις ερωτήσεις, όχι μόνο των συνδικάτων, αλλά όλων των ενδιαφερομένων, που βεβαίως άλλοι ενδιαφερομένοι είχαν άλλες ερωτήσεις από τα συνδικάτα. Δηλαδή το να παίρνουμε το κείμενο των άλλων όσο βάση του πακέτου δεν ισχύει. Ελπίζω λοιπόν σε λίγες μέρες όταν θα δείτε το πακέτο να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Μάλιστα δύο καλές ερωτήσεις και δύο καλές απαντήσεις. Καλύτερο από 7 κακές ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, έχω άλλη μια ερώτηση. Διμερείς αεροπορικές συμφωνίες. Πώς πάνε τα πράγματα. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Αζίαν προχωράει καλά. Αρμενία προχωράει καλά. Κόλπος πλην Εμμυράτων. Ε, ε, Περσικός κόλπος. Μια χαρά προχωράει. Και τώρα να ενθαρρύνουν να προτείνουμε νέε διαπραγματεύσει ε, λόγω αυτών των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Σχεδόν σεβαστήκατε, σχεδόν σεβαστήκατε το χρόνο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σμέλ Ερτούγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Ξεκινάω. Θα προσπαθήσω να κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις, ελπίζοντας ότι θα μας απαντήσετε πρώτον. Νομίζω ότι δεν είναι δική σας ευθύνη το ότι στα υψηλά κλιμάκια της ε, Κομισιόν τα ζητήματα της κινητικότητας είναι κάπως ε, σε δεύτερη μοίρα. Κυριακή μα είπατε ότι είναι σημαντικό θέμα, αλλά αν δούμε το πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν, τότε όπως τα βλέπω εγώ, η λέξη κινητικότητα εμφανίζεται μία φορά ως θέμα υποτεταγμένο στην ε, ανακοίνωση, τη σημαντική ανακοίνωση για τις χαμηλές εκπομπές. Τέλο, δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Π.χ. είδαμε την προηγούμενη περίοδο το πράσινο πακέτο για τις μεταφορές και κομισιόν είχε πει ότι μέχρι το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους θα έπρεπε να έχουν κατατηθεί όλα τα εθνικά σχέδια δράσης. Πρώτον, πρώτη ερώτηση. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι στιγμής 17 κράτη-μέλη έχουν αποστείλει κάτι πώς έχουν τα πράγματα συγκεκριμένα, ποιος δεν έχει στείλει, συγκεκριμένα χώρες θέλω και τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να εκπληρώσουν τα κράτη-μέλη της υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα επιτρέψατε μου μία διόρθωση. Μπορεί να είχε υποτιμηθεί να είχαν υποτιμηθεί οι μεταφορές στο πρόγραμμα του 2016, αλλά το 2017 κυριαρχεί στο πρόγραμμα εργασίας. Τα πράγματα βελτιώνονται και δεν μπορώ να πω ότι παραμελούμε πλέον τις μεταφορές. Ε, νομίζω περιλαμβάνεται σε όλες τις πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες ε, και στις ε, παγκόσμιε ε, και στις ε, πρωτοβουλίες ενιαία αγοράς και νομίζω οι μεταφορές σήμερα αφορούν το 21% των προϊόντων και 18% των υπηρεσιών που εξάγουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ακουγόμαστε σίγουρα. Τώρα, για τα εναλλακτικά καύσιμα. Έχετε δίκιο, υπήρξε κάποια καθαίριση. Απέστειλα προσωπικά μια επιστολή στα κράτη-μέλη πέρσι και 19 κράτη-μέλη έχουν απαντήσει. Ξεκινήσαμε με όλες τις άλλες χώρες σε διαδικασία παραβάση και άρα περιμένω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε απαντήσεις από όλα τα κράτη-μέλη και όπως ξέρετε ε, σκοπεύουμε να έχουμε πλήρη αναφορά σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. Ε, μπορώ να πω πως οι αποκλήσει είναι αρκετά μεγάλες, ε, οπότε υπάρχουν κάποιες ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Να ρωτήσω, να ρωτήσω επί του θέματος αυτού, ποιες εννέα χώρες μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει. Α, δεν τα ξέρω απ' έξω, μπορώ να στείλω μια λίστα. Ωραία. Ναι, όπως ε, είπε ο κύριος ε, Φάντεκαμπ, ε, υπάρχει η κοινωνική πτυχή. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάφορα προβλήματα, Βλέπουμε τις υποδομές στις κεντρικές χώρες, πώς υποφέρουν, ε, τι γίνεται στους αυτοκινητόδρομους με οδηγούς ε, φορτηγών και αυτοκινήτων. Γι' αυτό εξακολουθώ να έχω την ιδέα και την ελπίδα ότι υπάρχει κάποιο είδους αρχή, α, δεν με ενδιαφέρει το πώς θα λέγεται, η οποία θα συνεισφέρει από το επίπεδο των Βρυξελών έτσι ώστε να μην υπάρχει κοινωνικό dumping, να υπάρχει ανταγωνισμός και κυρίως να υπάρχει έλεγχος και επιβολή του νόμου. Το έχετε περιλάβει αυτό στο σχέδιο του οδικού πακέτου. Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα είναι να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες και να απλοποιηθούν. Γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα με το υφιστάμενο πλαίσιο. Φοβάμαι ότι υπονοείται κάποιο είδους ευρωπαϊκή αρχή. Πρώτα απ' όλα ακούσαμε την ε, σύσταση του Κοινοβουλίου κάποιων συναδέλφων σας. Βλέπουμε κατά πόσο μπορούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν επιτυχώς κανόνες. Εάν ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη ευρωπαϊκής επιβολής, οπωσδήποτε θα δράσουμε. Παρατηρούμε τώρα την εφαρμογή ε, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όχι μόνο τα κοινωνικά ζητήματα, το ζήτημα της απομάκρυνσης από τον άνθρακα κτλ. Και εάν οι εθνικές υπηρεσίε δεν είναι αρκετά επιτυχίες, θα προτείνουμε περαιτέρω βήματα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση του προγράμματός σας. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι ε, Δεκτώ αυτό το οποίο λέτε ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία και επιπροσθέτως ε, θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τους υφιστάμενους κανόνες. Δεν υποστηρίζουμε την επιπρόσθετη νομοθεσία επειδή δεν εφαρμόστηκε η ε, αρχική. Γιατί τελικά καταλήγουμε με όλο και περισσότερη νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Μία μικρή ανησυχία αναφέρατε το, στο πακέτο κινητικότητας το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα και των εκπομπών για τα φορτηγά. Σημαντικό, αλλά εμείς έχουμε μια ατζέντα για, την, για τις μεταφορές και έχουμε άλλες επιτροπές που λέγονται απασχόλησης και άλλοι λέγεται περιβάλλοντος. Ε, και πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε εδώ πέρα στον τομέα των μεταφορών και το τι μπορούμε να κάνουμε ε, από την πλευρά των μεταφορών, ανεξαρτήτως της καλής ε, συνεργασίας που έχουμε. για το θέμα της ασφάλειας ε, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, να πω κάτι πριν κάνω την ερώτησή μου. Θα ήταν χρήσιμο αν όλα τα κράτη-μέλη απαγόρευαν την χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Γιατί βλέπουμε κόσμο να μιλάει στο κινητό, να γράφει στο κινητό, να μην κοιτάει μπροστά του και πλέον είναι σημαντική αιτία ατυχημάτων ε, τα κινητά και έρχομαι άρα στον σιδηρόδρομο και αυτό το οποίο αναφέρατε με το through ticketing. Το έχουμε εδώ και χρόνια το θέμα και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει. Έχει γίνει στον τομέα της αεροπορίας εδώ και 40 χρόνια. Υπάρχουν εταιρείες, δεν διαφημίζω τώρα, αλλά μπορούμε να μπούμε στο διαδίκτυο, να βρούμε τέτοια ειστήρια ε, για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό το οποίο έχουμε, φοβάμαι, είναι ότι έχουμε ακόμα κάποια κατημελή με σιδηροδρομικές εταιρείε που δεν θέλουν να έρθουν στον 21ο αιώνα ε, ή να φέρουν τον καταναλωτή στον 21ο αιώνα. Θέλουν να έχουν ε, προτεραιότητα οι ίδιοι και δεν ε, εξετάζουν ακριβώς το πρόβλημα. Οπότε, για το πρώτο αυτό ζήτημα του through ticketing, τι θα κάνει και γι' αυτό η Κομισιόν. Είναι ζήτημα προστατευτισμού και οπωσδήποτε δεν το δέχεται η Επιτροπή μας. Λοιπόν, βοηθήστε με αν ξεχάσω κάποια ερώτηση. Άκουσα... Λοιπόν, με το ερώτημα με τα ειστήρια. Γνωρίζω το πρόβλημα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ε, ήδη εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμε με το πώς θα βρούμε μια στιβαρή αρχιτεκτονική για τις μεταφορές. Εννοώ αρχιτεκτονική δεδομένων για να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι οπωσδήποτε το μεγαλύτερο ζήτημα διατροπικών μεταφορών, όχι μόνο για τα τρένα, αλλά για όλα αυτά τα περιβάλλοντα. Θεωρώ ότι του χρόνου θα έχουμε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες σε όλες αυτές τις συζητήσεις ε, για να δούμε αν πρέπει να γίνει κάτι στο θέμα τυποποίησης στο νομοθετικό επίπεδο για να πρέπει να ενθαρρύνουμε τις εταιρείε ε, να αρχίσουν να συνεργάζονται. Ελπίζω λοιπόν να μας στηρίξετε κι εσείς. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Οι άλλες δύο ερωτήσεις ήταν, ε, σχόλια. Λοιπόν, μιλήσατε για προτάσεις για την αυθυλία και την αεροπορία. Και προφανώς τα αναμένουμε. Νομίζω ότι ε, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα δεν θέμε αλληλεπικάλυψη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ενώ πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχει ήδη συμμόρφωση με αυτά τα οποία λέει ο IMO. Και νομίζω ότι πηγαίνουν αρκετά καλά τα πράγματα στην ασφάλεια και σε άλλου τομεί, οπότε αναμένουμε να δούμε το τι θα προτείνεται με τις λοιπέ ε, προτάσεις για την αυτιλία. Και τέλος για την αεροπορία, είναι ηρωνικό, δηλαδή μιλάμε για έλεγχο και η τρίτη φάση τη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τους ε, ανοιχτούς ουρανούς. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τα ζητήματα ελέγχου και ιδιοκτησίας. Ε, οπότε είναι και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Αναφέρατε την ΙΑΖΑ. Ε, υπάρχει κάποια ερώτηση, κυρία Φώστερ, κάποτε. Και το τελευταίο θέμα, ε, η ερώτηση μου είναι αν συμφωνείτε ότι θα πρέπει να σταματήσει το χρονόμετρο για να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα εκπομπών για την αεροπορία για το μέλλον. Συμφωνείτε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, να απαντήσω. Κοιτάξτε, οι κατευθυντήριες γραμμές της 7 ε, Ιουνίου θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Κύριε Τενίτσικα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα ξεκινήσω με δύο απλές αφελείς ενδεχομένως ερωτήσεις. Οι δέσμοι μέτρων για την κινητικότητα είναι δέσμοι γιατί ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές προτάσεις ή υπάρχει πραγματικά μια εστερική συνοχή στις προτάσεις αυτές. Θέλουμε να έχουμε μία εσωτερική ισορροπημένη συνοχή, η οποία θα λάβει χώρα σε διάφορες φάσεις. Έχουμε ήδη μία εικόνα εκ των προτέρων, γι' αυτό το λόγο υποβάλλουμε εξ αρχής μία δέσμη μέτρων. Σε δύο φάσεις θα υποβληθούν οι προτάσεις αυτές, ήδη κάποιες από φέτος και κάποιες προτάσεις του χρόνου. Κατάλαβα καλά ότι στη φάση αυτή δεδομένου το ότι υπάρχει μια κοινωνική, περιβαλλοντική, ψηφιακή πτυχή, πτυχή εσωτερική αγορά, θα λέγατε λοιπόν ότι οι υπόλοιποι επίτροποι που είναι υπεύθυνοι για του τομεί αυτού ε, συμφωνούν μαζί σα, έχετε τη δική του συνένεση. Απάντηση καταφατική. Πολύ ωραία. Τότε συμφωνείτε μαζί μου λέγοντας ότι προκειμένου να φτάσουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν μια προσέγγιση δέσμης μέτρων, δηλαδή να υπάρχει παράλληλη προσέγγιση για όλες τις προτάσεις. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, συμφωνείτε ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα καταφέρουμε να, φτάξουμε, να φτάσουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα. Έχω δίκιο. Να σας απαντήσω λίγο εκτενέστερα αυτή τη φορά, λέει Επίτροπος θα δείτε ότι ορισμένες προτάσεις, νομοθετη... νομοθετικές προτάσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο, άλλες λιγότερο. Αν έχουμε όμως την κατάλληλη συνεργασία θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε συντονισμένα στα πλαίσια της δικής μου εντολής για το σύνολο της δέσμης μέτρων. Αν υποβληθεί όμως όλη αυτή η πρόταση αυτή ως δέσμη θα πρέπει να παραμείνει ως δέσμη, έτσι δεν είναι. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολλές διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με την αεροπορία. Μας είπατε τι περιμένουμε ήδη από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφική σας, αν θέλετε, προσέγγιση και πώς σας συνάδει με τις υπόλοιπες επιμέρους συμφωνίες που έχουμε στην αεροπορία. Ποια είναι, πώς συνάδει η γενικότερη προσέγγιση που έχουμε στην αεροπορία με τις διμερείς συμφωνίες. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση. Το 86 είναι ένα εργαλείο απλώς το οποίο χρησιμοποιούμε προκειμένου να σημειώνουμε πρόοδο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το εργαλείο αυτό συνάδει ιδιότερα για την αεροπορία. Είναι καλύτερα, αν θέλετε, προσαρμοσμένο στην αεροπορία. Στο παρελθόν είχαμε ένα άλλο μέσο το οποίο χρησιμοποίησαμε περισσότερο γενικότερα για το τομέα του εμπορίου. Με το νέο 868 όλες οι φάσεις των παραπώνων αναφέρονται ξεκάθαρα έχουμε την κατάλληλη διαχείριση, την κατάλληλη επεξεργασία κάθε φορά στο κατάλληλο επίπεδο προκειμένου να μπορούμε να σημειώνουμε πρόοδο και προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη αν θέλετε για κάθε καταγγελία. Μολονότι δημοσιεύτηκαν πάρα πολλά άρθρα, ακούστηκαν πάρα πολλές φήμες για το ότι δεν λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα με το νέο 868. Στα πλαίσια του νέου αυτού εργαλείου δεν έχει υποβληθεί καμία νέα καταγγελία. Πάντως με το νέο αυτό μέσο, με τη νέα αυτή οδηγία, σίγουρα θα έχουμε το κατάλληλο εργαλείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά από τα κράτη-μέλη όταν θεωρούμε ότι υπάρχει μία παρατυπία στα πλαίσια των αερομεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Επομένως, έχουμε μία συμπληρωματικότητα προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Μία ακόμα ερώτηση που έχει να κάνει με το ενιαίο αυτό εισιτήριο, το εισιτήριο κατευθείαν. Ήδη αναφερθήκατε σε αυτό. Θα λέγατε όμως ότι ανεξάρτητα της τυποποίησης, γιατί αυτό έχει προκύψει ως θέμα, και ανεξάρτητα της απαιτούμενης νομοθεσίας, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα σημεία συμφόρησης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι στα πλαίσια της δικής σας εντολής θα υποβληθεί επισήμως μια πρόταση προκειμένου το ενιαίο αυτό εισιτήριο, του εισιτήριο κατευθείαν να αποτελέσει τελικά πραγματικότητα. Από πλευρά επιβατών, ναι. Πολύ ωραία. Τελική τώρα ερώτηση. Τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τους δείκτες συνδεσιμότητας για την αεροπορία. Ενδεχομένω υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιεί δείκτες συνεκτικότητας. Κοιτάξτε, εμεί καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες για αυτό το δείκτη συνδεσιμότητας. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως συγκεκριμένε ημερομηνίε αυτή τη στιγμή για κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα. Έχω 13 ακόμα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε. Ναι, ξέρετε την απάντηση, δείτε λίγο το βλέπα μου. Η κυρία Κίλωνεν τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο, κύριε συνάδελφοι, κυρία Επίτροπο. Μια ερώτηση για την αεροπορία καταρχάς. Η πίστοση συνάπλωση αεροσκαφών, airport charting, θα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Και επόμενο, έρχομαι στο αυθενό προξεναλλακτικά καύση. Δύο σεμινάρια ε, προβλέπονταν για την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει, με εξέπληξε το γεγονός αυτό. Ότι δηλαδή ανταλλάσσουμε πολύ λίγες πληροφορίες, πολύ και πολύ λίγες καλές πρακτικές. Οι συναντήσεις αυτές που σας είπα τις προηγούμενες εβδομάδες, στα σεμινάρια αυτά, διαπίστωσα ότι κάνουμε τις ίδιες μελέτες. Ελέγχουμε τις ίδιες πληροφορίες. Όλα αυτά με χρήματα που προέρχονται από, το, από τον ενωσιακό προπολογισμό. τα ίδια πράγματα από διαφορετικές χώρες. Τι μπορείτε να κάνετε ώστε την ε, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, ιδίω στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και στον αεροπορικό τομέα και στον τομέα των οδικών μεταφορών, να μην χρειάζεται να δαπανώνται έτσι τα χρήματα των φραγμένων αλλά να δαπανώνται με πιο συνετό τρόπο, γιατί μετά λέμε δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Εγώ άρχισα να συνειδητοποιώ όμω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ότι δεν κάνουμε σωστή χρήση των κονδυλίων και ένα μικρό δωράκι. Δεν είναι το πόσιμο νερό βέβαια. Αλλά κάτι για τα απόβλητα. Θα ήθελα να είναι πιο πράσινη η, η στόλη. Green wash. Αυτό είναι αυτό που θέλω να υποστηρίξουμε. Θα ήθελα να ελέγξετε και με πολύ ανοιχτό μυαλό το που πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Να έχουμε δηλαδή καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά οι θάλασσες να είναι τόσο πολύ μολυσμένες. You, uh, if I very quickly, uh, Απάντηση. Airport charges, όχι charting, διορθώνει διερμηνέα ε, για τα αεροπορικά τέλη. Είναι, είμαστε σε διαβουλεύσεις και σε δύο εβδομάδες θα έχουμε ε, μια νέα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας δώσω μια ημερομηνία ως προς το τι θα προτείνουμε, αλλά τα συζητούμε, είναι μέρος ε, των διαβουλεύσεων και της στρατηγικής και θα δούμε τι θα προκύψει. Το δεύτερο για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται και είναι τα ίδια, αλλά σε διαφορετικές χώρες, ανταλλαγή προφών λοιπά, Πράγματι, είναι πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με καλύτερο συντονισμό και πραγματικά καταρρύπτουμε πολλά στεγανά, γκρεμίζουμε στεγανά από πλευράς μεταφορών. Έχω να σας μεταφέρω μια θετική εμπειρία Θέλουμε να επενδύουμε μία φορά μόνο. Έχουμε κοινοπραξίε τώρα στην αεροπορία και στους σιδηροδρόμους σεζαρ και Shift to Rail. Και πραγματικά φαίνεται ότι είναι πολύ καλό εργαλείο για καινοτομία, όχι για έρευνα ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να παραμείνει. Στην ακαδημαϊκή έρευνα, στα διάφορα ιδρύματα και τους κύκλους ανάπτυξης. Όμως φαίνεται ότι οι κοινοπραξίες καινοτομία είναι κάτι θετικό και θα συνεχίσω να το ενθαρρύνω και ελπίζουμε να έχουμε και κάποιες ακόμη κοινό πραξίες. Τους πράσινους τόλους. Σίγουρα θέλουμε να πρασινίσουν μεταφορές και ένα από τα πιο καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα ήταν ε, να έχουμε πιο οικολογικά πλοία, πιο οικολογικά σκάφη και σιγά σιγά δίνει καρπούς το project αυτό. Σίγουρα ένα θέμα το οποίο σε επίπεδο ναυτιλιακού οργανισμού μα απασχολεί ιδιαίτερα και βέβαια οποιαδήποτε υποστήριξη, ενθάρρυνση από τα κράτη-μέλη θα ήταν καλοδεχούμενη για να βρεθεί μια γενικότερη, μια παγκόσμια λύση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Ο επόμενος ομιλητής τώρα έχει το λόγο. Commissioner. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γιάκουμ Νταλούντα. Ο τομέας των μεταφορών πρέπει να χαρακτηρίζεται από πιο δίκαιο ανταγωνισμό, διότι αυτή τη στιγμή ευνοούνται σημαντικά και δυσανάλογα οι οδικές μεταφορές και το πληρώνουν το τίμημα, οι κοινωνίες με συμφόρηση, ε, με τη ρήπανση, με το κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου και βέβαια ε, υποβάθμιση και του συνδρομικού δικτύου. Για τα διόδια θα πρέπει η σχετική νομοθεσία να συμφωνεί με τη Συμφωνία των Παρισίων. Χιλιομετρικά θα πρέπει να υπολογίζεται τι με τον διοδίων. Είναι μια λύση, ισχύει σε κάποιε χώρε και στη δική μου τη χώρα, τη Σουηδία, σκεφτόμαστε να το εφαρμόσουμε. Γιατί να μην ισχύσει εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να έχουμε και ισότιμο ανταγωνισμό. Πώ ο τομέα των αδικών μεταφορών θα πληρώσει το μερίδιο που το αναλογίζει ό,τι αφορά το κόστος των ε, υποδομών και το εξωτερικό κόστος. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, αν επιτρέπετε. Το 2014 έως 2020, από πλευράς επενδύσεων, τονίζουμε τους σιδηροδρόμους, αυτό το, την αλλαγή παραδείγματος περιμένουμε να ολοκληρωθούν αυτά τα project, τη χρηματοδότηση όμως σε μεγαλύτερο βαθμό πηγαίνει στη συνολική συνδεσιμότητα τους ε, κρίκους αλήθειας που λείπουν και στους σιδηροδρόμους. Για το ERTMS χαίρομαι που στην τελευταία αναθεώρηση του σχεδίου δράση, το Δεκέμβριο πέρσι δηλαδή, ε, εγκρίναμε κάτι θετικά πράγματα. Πρέπει βέβαια να αρχίσουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν οι σιδηρόδρομοι. Δυστυχώ εκεί δεν βλέπουμε τι εξέλιξεις που θα επιθυμούσαμε όσον αφορά την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά ε, τα τέλη και τις διάφορες επιβαρύνσεις, ε, φυσικά και θα ε, διατυπώσουμε προτάσει για αλλαγέ το 2018. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε σε βάθο. Όλου του φόρου και όλε τι επιβαρύνσει για όλου του τρόπου μεταφορά, Ο κ. Κράμερ ξέρουμε ότι το υποστήριζε στεναρά, μας πίεσε και πράγματι πέρυσι αναλάβαμε αυτή την προσπάθεια και την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι θα δείτε με την ανάλυση μας ε, ότι θα ε, ξεκαθαρίσει και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για όλους τους τρόπους μεταφορών και για να έχουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Charging, road charging, sorry. Thank you. τα οδικά τέλη τώρα. Στα πλαίσια της δέσμης κινητικότητας έχουμε την Ευρωβινιέτα και κάποιες άλλες ψηφιακές λύσεις όσον αφορά τα οδικά τέλη που περιλαμβάνουν όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και στελεστές. Καλούμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι θα ισχύσει η αρχή ότι ο χρήστης πληρώνει, ότι ο ρηπαίνων πληρώνει και να χρησιμοποιηθούν οι νέοι αυτοί μηχανισμοί προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτά τα οδικά τέλη και τα τέλη που έχουν να κάνουν με την κυκλοφοριακή συμφόρηση ή με, τη, τα τέλη μόλυνσης ε, και το καθεξής. Και νομίζω ότι όντως τα τέλη τα οποία θα βασίζονται στην απόσταση θα είναι πολύ πιο δίκαια τέλη από το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα. Εμείς σε καμία περίπτωση όμως δεν επιβάλλουμε ένα σύστημα δικών τελών αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να κινηθούν προς αυτό το σύστημα που προτείνουμε εμείς για τα οδικά τέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με το προτινόμενο από εμά ευρωπαϊκό μοντέλο. Αυτό για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Περνά τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Πριν από χρόνια, όταν ήταν ε, νέοι οι γονεί μου, μπορούσαν να πάρουν ε, ένα τρένο από τη Στοκόλμη, να ξυπνήσουν την επόμενη μέρα στο Παρίσι, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ε, πόλη. Και αυτό γιατί βέβαια παίρνανε νυχτερινά τρένη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτά τα τρένα έχουν καταργηθεί και ότι η μόνη λύση που έχει πλέον κανεί να πάρει το αεροπλάνο για αυτέ τι μικρέ ή μεσαίε, αν θέλετε, αποστάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει, αν θέλετε, για να αναστρέψει την τάση αυτή, για να σώσει τα λίγα να απομείναντα νυχτερινά τρένα. Θα σας στενοχωρήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει να επέμβει αυτή τη στιγμή και να επηρεάσει τη δυναμική της αγοράς. Σωστό και θεμητό το ερώτημά σα για ποιο λόγο ορισμένε μορφέ υδροδρομικών μεταφορών δεν αναπτύσσονται τόσο σε άλλε μορφέ μεταφορών, όπω οι ε, οδικέ μεταφορέ ή άλλε μεταφορέ, που προσαρμόζονται πολύ περισσότερο στι ανάγκε κινητικότητα, πολύ περισσότερο τελικά από ό,τι στη σιδηρόδρομη. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε, πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτρομή, Επιτροπή προσπαθεί κάθε διδροδρομη δεν μπορουμε να εξισορροπήσει τα πράγματα και να ενθαρρύνει όλο και περισσότερο και την εναρμόνιση αλλά και τις επενδύσεις για του σιδηροδρόμου, Ξέρετε ότι καταφέραμε να αντικαταστήσουμε περίπου 11.000 εθνικού κανόνε με 400 ευρωπαϊκού κανόνε στα πλαίσια τη τέταρτη σιδηροδρομική δέσμη. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι τιμέ για τον εξοπλισμό το σιδηροδρομικό γίνονται πολύ πιο ανταγωνιστικέ και δημιουργούμε ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού όπου καταφέρνουμε και να προστατεύσουμε του επιβάτε, αλλά και να ανοίξουμε την αγορά σε περισσότερου φορεί εκμετάλλευσης οι οποίοι πολλέ φορέ είναι και πιο δυναμικοί και συνδυάζουν και και άλλες μορφές και άλλους τρόπους μεταφορών. Και βέβαια προσβλέπω και στις δικές σας ε, τις προτάσεις για να δω τι κενά θα μπορούσαμε να καλύψουμε. Το ζήτημα της φορολόγησης είναι κάτι το οποίο είχε θίξει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το έχουμε λάβει υπόψη μας, αλλά περιμένουμε από εσά και άλλες προτάσεις για να καταφέρουμε να τονώσουμε περισσότερο το σιδηροδρομικό κλάδο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω. Κοιτάξτε, στο θέμα των φορτηγών που έχουν περισσότερα ατυχήματα. Μα βεβαίω αυτό το οποίο προτείνετε δεν θα αλλάξει την κατάσταση γιατί υπάρχουν τα κενά στην ε, νομοθεσία περί καμποτάζ και υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπων με ελάχιστα λεφτά και ε, το μόνο που απομένει στους οδηγούς είναι να ε, το ρίξουν στο πιωτή. Συχνά στην Σουηδία πιάνουν οδηγούς πιωμένου και πρέπει να δούμε το πρόβλημα του καμποτάζ. Εκείνη η ρίζα του ζητήματος και ε, έχουν ακόμα και πλαστά διπλώματα οδήγησης ε, που βρίσκουμε. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν σκέφτεται να φτιάξει μια ε, διεθνή βάση δεδομένων ή διπλωμάτων ή να υπάρχει δυνατότητα στην αστυνομία να ελέγξει αν γνήσει τα διπλώματα. Ναι, ναι, Πρώτα απ' όλα γνωρίζω πολύ καλά τις ε, συνθήκες, έχω πάει με τους δαλικέρδες, έχω πάει με την τροχέα στα μπλόκα. Εγώ βεβαίως εντάξει αυτό δεν έχω δει ούτε το 1% των όσων συμβαίνουν, αλλά πήρα μια ιδέα. Ε, υπάρχουν και αντιεπαγγελματικές ε, συνθήκες, τις οποίες υφίστανται πολλοί οδηγοί. Γι' αυτό ακριβώς το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα κοιτάμε το καμποτάζ, τις συνθήκες εργασίας. Ένα από τα πιο προβληματικά σημεία που συμβαίνουν στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά οι εταιρείε γραμματοκιβώτια. Για το καμποτάζ, πρέπει να πω ξεκάθαρα. Διαβουλευόμαστε με τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν αλλάζουμε τους κανόνες της αγοράς με την έννοια να ανοίξει, να κλείσει η αγορά αλλά θα προτείνουμε κάτι το οποίο θα μπορεί να επιβληθεί γιατί υπήρχε απέτηση από την αγορά να έχουμε κανόνες οι οποίοι θα επιβάλλονται και θα ελέγχονται εύκολα. Και αυτό πάει χέρι με χέρι με τη βελτίωση των συνδικών εργασίας ε, όσον αφορά τους χρόνους ανάπαυσης ε, και βεβαίως ε, τις αμοιβέ. Αυτά πάνε μαζί. Κοινωνικά ζητήματα με ζητήματα αγοράς. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να τα βλέπουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω πως ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώ ε, τις ψεύτικες έδρες και πηγαίνουμε προς ένα μοντέλο το οποίο θα απαιτεί από τις εταιρείε ε, εκεί όπου έχουν έδρα να επιτελούν και το, το κύριο έργο τους το, το διοικητικό. Αλλά τα περισσότερα λεπτομέρειες ε, προσεχώς. Ε, ευχαριστώ. Οι οδηγοί που πίνουν. Το πρόβλημα με αυτού είναι το εξή. Έχουμε διάφορα όρια αλκοολεμίας ε, στις διάφορες χώρες. Και αυτό προκαλεί προβλήματα. Ε, είχαμε την Υπουργό στην Σουηδία των Σοσιαλδημοκρατών που πήγε στη Δανία με το αυτοκίνητο. Νόμιζε ότι ήταν εντό του ορίου γιατί είναι ψηλότερο στη Δανία αλλά μετά τη κάνανε αλκοτέστ στην ε, Σουηδία και την συλλάβανε. Μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ένα κοινό όριο αλκοολεμίας για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Γιατί ο κόσμος πάει σε άλλη χώρα, νομίζει ότι ξέρει τα όρια και τελικά βρίσκεται... Uh, Έχετε δίκιο. Πράγματι, διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες. Και είναι εθνική αρμοδιότητα. Και αυτό ισχύει και για τα όρια του αλκοόλ στο αίμα. Εγώ ευχαριστώ να συζητήσω το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι στο πακέτο δικής ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει με τους ε, συντονιστές ε, και τώρα περνάμε στον επόμενο γύρο. Ε, δυστυχώς όμως, αντί για τρία λεπτά, γιατί θα περάσουμε όλη μας τη μέρα εδώ, αν το αφήσω, θα έχετε δύο λεπτά ο καθένας και θα ξεκινήσουμε την κυρία Λουκασένσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η πρώτη είναι η εξής. Είστε υπέρ ε, της πρότασης ε, να καλύπτονται οι μεταφορές από την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Εάν ναι, γιατί. Εάν όχι, τι θα κάνετε για να μην ε, περιληφθεί στην ε, οδηγία περί απόσπασης ε, ο τομέας των μεταφορών. Έχουν την εντύπωση ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης πολλοί, επιτροποί θέλουν να, πολλοί συνάδελφοι με θέλουν να συμπεριληφθεί. Δεύτερον, θα ήθελα για μια συγκεκριμένη απάντηση. Διαδικασίες ε, επί παραβάση που έχουν ξεκινήσει για τον βασικό μισθό στη Γερμανία. Πού βρισκόμαστε. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια στάσιμότητα, δεν υπάρχει κάποια πρόοδος. Έχουμε κολλήσει. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Η διαδικασία αυτή γιατί ξεκίνησε για τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία και τώρα βρίσκονται στο επίπεδο της επίσημης ε, επιστολής. Ε, βλέποντας πως, ε, πόσα κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν κάποια εθνική δραστηριότητα, είπαμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δεύτερη ερώτηση για την απόσπαση εργαζομένων και τη σχετική οδηγία. Βεβαίως η οδηγία αυτή ε, ισχύει για όλους τους κλάδους ε, και τις οδικές μεταφορές αλλά νομίζω και άλλοι το έχουν αναγνωρίσει και η συναδελφός μου η κυρία Ταΐσεν ότι θα αναγνωρίσουμε το ειδικό καθεστώς των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούση Άντρισον, για δύο λεπτά. Thank you. Just a of um, Ευχαριστώ. Κάνω δύο ερωτήματα σε σχέση με το σιδηρόδρομο κυρίως, όχι αποκλειστικά. Η μετατόπιση προς το σιδηρόδρομο, shift to rail, καλή πρωτοβουλία και ελπίζω να έχουμε και δεύτερο τέτοιο πακέτο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πώς έχει η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε και τόσο μεγάλη μετατόπιση ε, από πιο επιζήμιες για το περιβάλλον ε, μορφές μεταφορών, ε, τι θα κάνετε, ιδίως ότι αφορά το πακέτο κινητικότητας, για να αναγνωρίσετε το αυτό το γεγονός και σε σχέση με όσα είπαν οι συνάδελφοί μου, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, οδικές εμπορευματικές μεταφορές, 75% μερίδιο ακόμη. Δεν αρκεί λοιπόν η πρόοδος. Ε, και είχαμε στόχους ε, στη Λευκή Βουλή 2011 που δεν τους έχουμε πετύχει ακόμη. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα στόχο ε, ή μια πρωτοβουλία για τις εμπορευματικές μεταφορές σε σχέση ε, με το ΣΕΦ και άλλες χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως και με το Shift to Rail. Σταματώ εδώ γιατί έχω κι άλλο ένα που θέλω να ρωτήσω μετά. Απάντηση πολύ γρήγορα. Το φθινόπωρο σας είπα. Θα έχουμε τη συνδυασμένη πρόταση της μεταφορές και ελπίζω να αυξηθεί το ποσοστό. Σίγουρα πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ε, ζητήματα για τους ε, σιδηρόδρομου. Να πάμε ε, από το σημείο στο σημείο Β με ένα φορτηγό είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά χρειάζεται λογική διαδρόμου για το σιδηρόδρομο. Γι' αυτό και εστιάζουμε τόσο πολύ στους διαδρόμους. Αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση διαδρόμου τέλος πάντων κυρίως για κάποια τμήματα ολοκληρωμένα. Δεν θέλουμε να έχουμε κατακαιρματισμένους διαδρόμους και οι συντονιστές μας νομίζω ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή πρόταση την οποία επεξεργάζονται. Ευχαριστώ. Άντερσον. Στηρίζω τον κύριο Ντελούντ και έχω την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση για τα νυχτερινά τρένα. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στις αγορές, αλλά θα πρέπει να δώσουμε στους καταναλωτές επιλογές ε, και για το περιβάλλον. Επειδή δεν υπάρχουν πάγια έξοδα, τα ε, λεωφορεία είναι πολύ φθηνά για το Uber ε, και για τη συνεργατική οικονομία στην ΙΜΚΟ. Εγκρίναμε μια έκθεση σήμερα. Δεν έλεγε ονόματα βέβαια, αλλά έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ ανησυχίε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία για τη συνεργατική οικονομία. Η δική σα γάμα τι κάνει. Ιδίω ό,τι αυτό το πακέτο κινητικότητα και επειδή θα έπρεπε να είχαμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Ότι δεν πρέπει αυτό να θεωρούνται μεταφορικέ υπηρεσίε. Η απάντηση δεν είναι μέρο ε, του πακέτου κινητικότητα. Πρόεδρο. Λοιπόν, πρέπει να παίξετε το παιχνίδι σωστά. Δύο λεπτά είχε το καθένας για να απαντάει και επίτροπος όμως μέσα σε αυτά τα δύο λεπτά. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά τα δύο λεπτά είναι δύο λεπτά. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ, έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη αφορά τα ασφαλή πάρκινγκ αποτελούν για, σε αυτοκινητόδρομους, αποτελούν τμήμα του πακέτου κινητικότητας. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίε οδηγοί που αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα και τους απειλούν, γίνονται διαρρήξεις στα οχήματα. Οπότε τι θα γίνει με, αν θα περιλάβετε ασφαλείς χώρους στάθμευσης. Δεύτερον, στους κανόνες ε, περί καμποτάζ ε, ε, αναφέρεται σε μία περίπτωση 7 ετών μπορούν να γίνουν ε, τρία ταξίδια, εντός, ε, τρία ταξίδια εσωτερικού. Και μετά. Ερώτηση. Τι θα κάνετε και με τον μισθό, το βασικό μισθό της ε, χώρας η οποία φιλοξενεί. Που θα αντικατασταθεί πλέον από το βασικό μισθό της ε, χώρας προέλευσης. Σας ευχαριστώ. Um, first of all, uh, parking... Καταρχάς, όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης, προσπαθούμε όντως να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους υπουργού από τα κράτη-μέλη ότι υπάρχει χρηματοδότηση από τον ΣΕΦ αυτή τη στιγμή για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης και ξέρουμε ότι πολλοί οδηγοί φορτηγών μας λένε ότι οι ασφαλιστικέ εταιρείες δεν ασφαλίζουν τα φορτηγά τους αν δεν κοιμούνται μέσα σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε κάθε φορά ότι ε, όταν προβλέπεται στάθμευση και χώρο στάθμευσης και όταν οι οδηγοί τελικά πρέπει να ξεκουραστούν και να πάνε σε κάποιο ξενοδοχείο, αρκεί να προβλέπεται αυτό βέβαια και να παρέχεται από την εργοδότη, τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν πώς μπορούν να διασφαλίσουν τους χώρους στάθμευσης και ήδη τώρα προβλέπεται χρηματοδότηση για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης. Προβλέπεται στα πλαίσια του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα το καμποτάζ, τη δεύτερη ερώτησή σας, επί του παρόντος είναι ανά αριθμό δράσεων και όχι σε χρονική περίοδο, δεν διαρθρώνται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά σκεφτόμαστε για αυτό το οποίο είπατε εσείς. Να έχουμε δηλαδή καμποτάζ το οποίο να διαμορφώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε ο κύριο Κούν λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη για την απάντηση αυτή. Ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Ευρωβινιέτα για τα τέλη, εναρμόνιση των δύο Ε, δεν εννοώ το ύψος των διοδίων, αλλά στο σύστημα να μην έχουμε όλα αυτά τα μηχανηματάκια που αγοράζει ο καθένα σε κάθε χώρα. Είναι γεμάτα τα παρμπρίζ από αυτά τα μηχανηματάκια. Δεν βλέπει ο οδηγός. Οπότε θα μπορούσε η Κομισιόν να ζητήσει να γίνει ένα, μια κοινοπραξία από τους μεγάλους Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία να έχουμε ένα σύστημα έτσι ώστε να μπορούν να περνούν τα σύνορα χωρίς να γίνεται ε, αυτή η δουλειά κάθε φορά που σταματάνε στα σύνορα και στα τελωνία. Ναι, ε, ενδιαφέρον το όραμά σας, συμφωνώ, η Κομισιόν θα προετοιμάσει μια πρόταση η οποία θα δώσει την δυνατότητα να υπάρξουν κάποιες ψηφιακές ε, πανευρωπαϊκές λύσεις, κάτι παρόμοιο με την αρχή ε, της ε, περιαγωγής στην τηλεφωνία. Αν θέλουν να συνεργαστούν οι εταιρείες, να συνεργαστούν. Υπάρχουν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης και μπορεί να υπάρξει και χρηματοδότηση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι. Δεν προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια τεχνολογία. Ευχαριστούμε, Ροβαντόλεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, να αναφερθώ στην δέσμη οδικών μεταφορών και κυρίως στην κοινωνική πτυχή, την οποία αναφέρατε και εσείς στην παρέμβασή σας. Είπατε και εσείς ότι όσον αφορά την οδική ασφάλεια έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και αυτό έχει να κάνει πολύ συχνά με τις συνθήκες εργασίας των οδηγών φορτηγών, για παράδειγμα. Αναφερθήκατε σε διάφορες φήμες, οι οποίες είπατε ήταν αβάσιμες. Και αναφερθήκατε επίσης στην μείωση της εβδομαδιαίας διάρκειας ανάπαυσης για τους οδηγούς. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε σήμερα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποβάλλετε πρόταση η οποία να συνάδει με τις φήμες οι οποίες ακούσαμε και η οποία ανησυχεί ιδιαίτερα τις δικαλιστικές οργανώσεις. Πρέπει επίσης να πούμε ότι το σύνολο των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σε δήλωση στη Βαρσοβία στις αρχές Απριλίου συμφώνησαν ότι είτε πρόκειται για χώρες της Κεντρικής ή της Ανατολικής Ευρώπης θέλουν να πετύχουν ένα νέο ευρωπαϊκό τέτοιο σύστημα. Μπορείτε λοιπόν εσείς να με σήμερα ότι θα υπάρξει μια μηνιαία χρονική διάρκεια όσον αφορά την άπαυση και θα συνεχίσει να υπάρχει μια εβδομαδία διάρκεια. 45 ώρες την εβδομάδα θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η διάταξη. Δεν είμαι πάντως πεπισμένη ότι με την πρόταση αυτή πραγματικά διασφαλίζεται την οδική ασφάλεια. Δεν είμαι πεπισμένη ότι 45 ώρες αυτές ανάπαυσης φτάνουν. Γιατί μιλάμε για ποιο είδος ακριβώς ανάπαυσης, τι είδους καμποτάζει τελευταία ανάλυση. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα συμπαγές, μια συμπαγή δέσμη μέτρων όπου να υπάρχει και αυτή η κοινωνική πτυχή και να μην υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην κοινωνική πτυχή, την περιβαλλοντική πτυχή, τι υπόλοιπε πτυχέ. Θα ήθελα να ασχοληθούμε επισταμένα με το ζήτημα τη οδική ασφάλεια και να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Απάντηση. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο, χρό... ο προβλεπόμενο χρόνο ανάπαυση εξακολουθεί να ισχύει. Πρόεδρος, ας συνεχίσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, τηρήστε το χρόνο αγόρευσης. Η κυρία Αϊούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Ήθελα απλώς να αφαιρθώ στο ζήτημα του 49% όσον αφορά τις ξένες οργανώσεις που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Το 2016 είπατε ότι ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιες διαπραγματεύσεις, Γαλλία, Γερμανία συγκεκριμένα, με χώρες του Περσικού κόλπου, προκειμένου να μην υπάρχει έντονη επέμβαση των χωρών αυτών του Περσικού κόλπου στις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες, γιατί ξέρετε ότι έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό πολλές φορές από τις εταιρείες αυτές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Έχουμε πρακτικές κοινωνικού dumping, για παράδειγμα, από τις ξένες αυτές αεροπορικές εταιρείες όταν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, για παράδειγμα, ευρωπαϊκών εταιριών. Πέρα όμω από τι επικρίσεις αυτέ που ακούστηκαν υπάρχουν και κάποιε μελέτε σύμφωνα με τι οποίε ο αθέμητο αυτός ανταγωνισμό των εξοκοινωτικών αυτών εταιριών με τι μεθόδου αυτέ, για παράδειγμα του κοινωνικού ντάμπινγκ έχουν πολύ δυσμενεί συνέπειε. Έχουμε όχι μόνο κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά το κοινωνικό αυτό ντάμπινγκ απλώνεται όλο και περισσότερο και παρισφρεί στι ίδιε τι πρακτικέ των ευρωπαϊκών αερομεταφορών μετά από τις διαπραγματεύσεις αυτές, πολλές φορές ήρθαν ακόμα σε εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια συγκεκριμένη εντολή για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό τομέα αερομεταφορών και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν αυτό το περιθώριο του 49% μπορεί αυτή τη στιγμή να εξακολουθήσει να ισχύει όσον αφορά δηλαδή τον έλεγχο που έχουν ξένες εταιρείες προς ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι το περιθώριο αυτό, το ποσοστό αυτό, δίνει τις, τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων. Ξέρετε ότι εμείς ε, στην Αλιτάλια, για παράδειγμα στην Ιταλία, ένα 49% ανήκει στην Etihad, που είναι ξένη εταιρεία. Εσείς προβλέπετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρρύψετε αν θέλετε το ποσοστό αυτό, να ξαναδείτε και να θεωρήσετε το ποσοστό του 49% όσον αφορά την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου στι Ευρωπαϊκέ Εταιρείε. Η επίτροπο έχει το λόγο και σας παρακαλώ πολύ να στηρίσουμε όλοι το χρόνο αγόρευσης. Κοιτάξτε, εμεί μόνο κατευθυντήριες γραμμές δίνουμε. Παράλληλα όμως κάνουμε και εμείς μία ανάλυση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αερομεταφορών βάσει της δικής σας πρότασης και όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση αυτή θα δούμε αν θα πρέπει να προταθεί περαιτέρω νομοθεσία ή όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κράμερ για δύο λεπτά. Μιλήσατε διόδια τα οποία θα βασίζονται στην απόσταση ε, για τους αλλοδαπούς οδαγούς η Γερμανία όμως έχει ακριβώς το αντίθετο και το δέχεται η Κομισιόν. Γιατί κύριε Κράμερ εσείς ξέρετε περισσότερα όπω ξέρω εγώ η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί η Κομισιόν ήταν σαφής μέχρι να δημοσιευτεί ο νόμος δεν θα δημοσιεύσουμε μόλις δημοσιευτεί θα σχολιάσουμε. Ταυτόχρονα θα είμαστε σαφείς ε, στην επικοινωνία για να δούμε τι μορφή θα πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, άρα αν παραμείνει το γερμανικό σχέδιο, η Κομισιόν θα πει όχι, γιατί δεν εξαρτάται από την απόσταση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι βινιέτε είναι εντάξει, αλλά όταν περάσει ο νόμος θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και όλα τα συστήματα θα αντικατασταθούν από ένα ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Είχαμε διαβουλεύσεις ήδη με ενδιαφερόμενους, ε, με τους ιδιοκτήτες ε, των συστημάτων και τώρα προσπαθούμε να δούμε ποια θα είναι μια λογική μεταβατική περίοδος. Μιλάμε ναι, για 25.000 νεκρούς από τροχιά. Έχουμε 400.000 νεκρούς από την ρήπανση της ατμόσφαιρας. Ακόμα και αν μειωθεί κατά 5% δεν είναι, είναι πιο είναι 25 φορές πιο βλαβερό ε, από το χειρότερο δίζελ. Γιατί δεν το απαγορεύετε. Κοιτάξτε, το να το απαγορεύσουμε σημαίνει ε, βλάβη σε πολλούς κλάδους. Ε, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα, ειδικά ε, τα ανανεώσιμα τα οποία στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να συγχρηματοδοτούμε, αλλά δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρώτα πηγαίνουμε στον τελικό χρήστη και τώρα πάμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πάμε και στην παραγωγή της ενέργειας με μαζούτ. Γεγονό είναι πως αυτή τη στιγμή οι μεταφορές κατά 93% βασίζονται στο πετρέλαιο. Κύριε Κώσου, έχετε τον λόγο. Κυρία Επίτροπε, μας μπερδέψατε λίγο. Μιλήσατε για ένα νέο πλαίσιο οδικής ασφάλειας το 2018. Τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, κατάλαβα καλά, είπατε πως ε, στο πλαίσιο της οδηγίας περί απόσπασης θα υπάρξει συγκεκριμένο κομμάτι για τις μεταφορές. Ισχύει αυτό? Ναι. Είναι η απάντηση. Και τι κρύβεται από το νέο πλαίσιο δικής ασφάλειας. Ε, δεν μου απαντήσατε στην πρώτη ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι είχαμε αυτή την δήλωση που υπογράφηκε στη Μάλτα από τα 28 κράτη-μέλη και όχι μόνο αυτό, είχαμε και τους εκπροσώπους της Ανατολικής Γειτονίας και των Βαλκανικών χωρών που επίσης έδειξαν ακριβώς ε, αφοσίωση στον να βελτιωθεί ασφάλεια και να πέσουν τα στατιστικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε πού και πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες υποδομών, το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η ζώνη, αλκοόλ, ε, ναρκωτικά και ταχύτητα. Και ελπίζουμε ε, αυστηρότερους κανόνες και επιβολή να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Συγκεντρώνουμε στοιχεία και χαίρομαι που επιτέλους μπορούμε να δούμε ποιος προκαλεί τα ατυχήματα, ποιος προκαλεί τα θανατηφόρα ατυχήματα, άνα χώρα, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι και τώρα από κοινού με τους υπουργούς ε, θα ρίνουμε τις εθνικές αρχές να δράσουν πιο σοβαρά. Κάτι άλλο το οποίο θα βοηθήσει είναι η συγχρηματοδότηση και η οδική ασφάλεια θα περιληφθεί σε αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μιλήσαμε, λέει κυρία Ταπαρδέλ, για σημαντικά στήματα δικαία η ασφάλεια, κοινωνικά δικαιώματα και το καθεξής. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω το ερώτημα των συναδέλφων. Είναι διαφορετικέ οι νομοθεσίε μεταξύ των κρατών μελών, άρα διαφορετικέ πολλέ φορέ και οι ερμηνείε περί τη εφαρμογή τη νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν καλό να έχουμε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τι Οδικέ Μεταφορέ. Μιλάμε για πολιτική υποστήριξη είναι ένας οργανισμός ε, που τρεις φορές το Κοινοβούλιο ε, ε, βρήκε υποστήριξη στην Επιτροπή Μεταφορών. Είχαμε την έκθεση για τα κοινωνικά θέματα. Είχαμε και ένα ψήφισμα για τις οδικές μεταφορές που τα ανέφερε. Θα ήθελα λοιπόν να το λάβετε υπόψη. Είναι μια πρόταση του Κοινοβουλίου με μεγάλη υποστήριξη. Έχουμε τόσους άλλους εκτελεστικούς οργανισμούς εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και για να σας αφήσω και χρόνο για να απαντήσετε, ήθελα, θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στις γυναίκες στις μεταφορές. Πολλές είναι οι γυναίκες στην Επιτροπή μας, βλέπετε ότι μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Τι γίνεται όμως με τον τομέα των μεταφορών. Το έχουμε θέσει το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί τάξη στα δράση και να διατυπωθούν νομοθετικέ προτάσει για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών ε, στη βιομηχανία των μεταφορών. Έχετε κάποια τέτοια πρόθεση. Ευχαριστώ. Απάντηση να ξεκινήσω από το τέλο. Νομίζω ότι προωθούμε ήδη από τώρα την ισότητα στι μεταφορέ και προσπαθώ να μην ε, μπω σε λεπτομέρειε, αλλά τέλο πάντων πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα που και άνδρες ε, θα καταλάβουν και θα νιώσουν ότι χρειάζεται να ε, υποστηριχθούν και αυτοί, ε, ώστε να υπάρχει ισότητα. Εμείς προσπαθούμε να ισορροπούμε μεταξύ των δύο φύλων και θέλουμε να ισορροπήσουμε και στη δική μου υπηρεσία, στη ΓΑΜΑ στο δικό μου πολιτικό γραφείο, θέλουμε να έχουμε την εις εκπροσώπηση των δύο φύλων και υπάρχουν ε, και προτάσεις επίσης για τις μεταφορές, θα τις ε, ακολουθήσουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν είναι ευνοϊκέ οι συνθήκε, θα έρθουν και γυναίκε. Αυτό ε, αυτή τη στιγμή μα απασχολεί, οι συνθήκε. Ευχαριστώ κύριο Λουί Δεγκράντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. ασφάλεια στην αεροπορία. Είμαι εισηγητής της έκθεσης ε, για τον εξοπλισμό ασφάλειας ε, στα αεροσκάφη. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, άλλοτε έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, άλλοτε μεγάλη ατολμία. Εσείς έχετε δίκιο στην Κομισιόν και θα πρέπει να δώσουμε μάχη ή ε, αντιθέτως θα πρέπει να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη ε, για να γίνει πιο ελκυστικό αυτό το νέο σύστημα και πρέπει να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις, να αλλάξετε κάποια πράγματα. Δεν καταλάβετε την ερώτηση. Well, I will just make a quick comment. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω στα σχόλιά σας. Εμείς συνεργαζόμαστε. Έχουμε και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τα θέματα ασφάλειας. King. Ο Επίτροπος Κίνγκ λοιπόν που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά συνεργαζόμαστε και αναλύουμε το πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ε, και την ασφάλεια της αεροπορίας αλλά και την ασφάλεια των αεροδρομίων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις που αποκλίνουν μεταξύ του, αλλά η ανάλυση θα μας δώσει, πιστεύω, όλα τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις προκλήσεις και όλα τα άλλα στοιχεία πρέπει να λέμε υπόψη. Και για το άλλο θέμα που αναφέρατε, συνεργαζόμαστε με τον Επιτροπό και θα δούμε ε, τι ε, πρέπει να γίνει για να έχουμε μια πολύ ξεκαθαρή θέση ό,τι αφορά την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Εγώ είπα ότι πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, ε, έχει δίκιο, όμως τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τα πράγματα με κινησμό, ενώ βλέπουμε τις επιθέσεις από την τρομοκρατία. Θα πρέπει να δώσουμε τους απαραίτητους πόρους για να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην αεροπορία. Ναι, να συνεργαστούμε, λέει η Επίτροπος. Πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και να έρθουν και τα κράτη-μέλη μαζί μας. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, όσον αφορά τον καποτάζ, θα το δούμε αυτό στο πακέτο της 31ης Μαΐου και θα έχουμε εδώ πέρα την περίοδο των τριών ημερών, γιατί κάτι τέτοιο ακούστηκε. Έπειτα, υπάρχει και υποχρέωση ανάπαυσης εκτός φορτηγού, το οποίο είπατε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Καθότι όμως θα αυξαθούν όλο και περισσότερο οι μεταφορές, καθώς επίσης και οι επιβάτες. Θα προβλεφθεί εδώ πέρα κάποια αλλαγή και περισσότερες επενδύσεις. Έπειτα, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες λύσεις προβλέπει προκειμένου αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η απάντηση είναι θετική, καταφατική για το καποντάζ. Όντως αποτελεί τμήμα του, της δέσμης μέτρων της 31ης Μαΐου. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε, όπως σας είπα, μια πρόταση που θα βασίζεται στη χρονική διάρκεια. Μπορείτε να επαναλάβετε το δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ πολύ. Ναι, προβλέπονται εδώ πέρα τρεις μέρες με, χωρίς να υπάρχει κανένα όριο για τις αναλήψεις που θα γίνονται. Δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα, λέει η Επίτροπος. Τελευταία ερώτηση. Ε, ένα ερώτημα όμως ακόμα, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την εθνική κρατική υποστήριξη θα υπάρχει ως προς κρατικές ενισχύσεις με καλύτερη ευελιξία. Κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με τι όμως ακριβώς, ρωτάει η Επίτροπος, όσον αφορά τις επενδύσεις για τη λειτουργία των αεροδρομίων. Όχι, όχι, δεν προβλέπετε τίποτα τέτοιο. Και ένα ακόμα ερώτημα όσον αφορά τις διατάξεις εκείνες για τα αεροπορικά σλότ και τα δικαιώματα των επιβατών που υπάρχει μπλοκάρισμα από ό,τι φαίνεται στο Συμβούλιο. Τι θα κάνετε με αυτά. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα διπλωματικής φύσης. Επί του παρόντος εμείς συνεχίζουμε τις διπλωματικές μας διαπραγματεύσεις αλλά ξέρετε ότι θα πρέπει να επιληθεί πρώτα και η διένεξη που έχει προκύψει μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας για το Γιβραλτάρ. Αν δεν επιληθεί η διένεξη αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γενικότερα στο φάκελο αυτό. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Κυρία Κούν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε όσον αφορά τον τομέα των αερομεταφορών και κυρίως όσον αφορά τις απεργίες των ελεκτών ενέργειας κυκλοφορίας. Από το 2010, 2,5 εκατομμύρια επιβάτες δεν έχουν καταφέρει πολλές φορές να ταξιδέψουν εξαιτία απεργίας των ελεκτών ενέργειας κυκλοφορίας. Το 2016 σπάσαμε κάθε ρεκόρ, γίνανε 22 διαφορετικές απεργίες στην Ευρώπη, 41 μέρες απεργίας και πάρα πολλοί ήταν οι επιβάτε αυτοί οι οποίοι επηρεάστηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια στρατηγική για τι αερομεταφορέ μετά την ανακοίνωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σιλέσκα ήταν ο εισηγητή μας και έχουμε και μία πρόταση για τους αεροδιαδρόμους, αν θέλετε αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Σαφώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να απεργεί, αλλά όταν έχει τέτοιες επιπτώσεις και στις χώρες μας και στις γειτονικές χώρες θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να διευκολύνετε τις μεταφορές, τις διασυνδέσεις και επίσης να μην υπάρχουν τι επιπτώσεις στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, στην ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου θα καλύψουμε και το ζήτημα αυτό, λέει η Επίτροπος, όπου θα εξηγήσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επί του παρόντος αυτό μπορώ να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και με όλες τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Προωθούμε την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια κάποια ευαισθητοποίηση και να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες, οι οποίες μιλούν από μόνες τους, θεωρώ, και θα μας οδηγήσουν τελικά στο να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία λύση. Το ζήτημα αυτό θα το καλύψουμε πάντως στην εκείνο 7 7η Ιουνίου. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε η Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Τηρήσατε το χρόνο αγόρευσης. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει τώρα, από εδώ και πέρα, θεωρώ να εγκρίνουμε τη μέθοδο αυτή ανταλλαγής απόψεων. Κυρία Άντερσον, κυρία Ιούτο, ξέρω ότι υπάρχει πολύ λίγος χρόνος ομιλίας, επομένως σας καλώ, εφόσον έχετε και άλλες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, να σας αποστείλετε γραπτό στην κυρία Επίτροπο και όσοι δεν κατάφεραν να πάρουν το λόγο, ας υποβάλουν και αυτοί μέσω email γραπτό στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους και θα απαντήσει προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι η ανταλλαγή αυτή απόψεων δεν είναι πάντα πάρα πολύ εύκολη. Σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων, καταγράψατε τις παρατηρήσεις μας και στις 19 Ιουνίου θα είμαστε σε θέση να επικεντρωθούμε περισσότερο στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήρθατε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και σε κάθε περίπτωση ελπίζω ότι καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό για όλα αυτά τα σημεία. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τη σειρά μου, λέει Επίτροπος, και κάθε φορά έχω την εντύπωση ότι περνάω από ακρόαση όταν έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ πάντω για τη δυνατότητα που μου δώσετε να πάρω το λόγο εδώ σήμερα. Ευχαριστώ.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

Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να βγουν από την αίθουσα χωρίς να κάνουν όμως τόρυβο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης «Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων». Η συγγήτρια είναι η κυρία Λούση Άντερσον. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο. Θα ακούσουμε συνέχεια τους σκιώδεις συγγητές ή άλλα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Και στο τέλος της συζήτησης θα καλέσω τον εκπρόσωπο, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να απαντήσει στο σύνολο των ερωτήσεων. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο. Thank you. And I'll try not to get told off. Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να μην μου κάνετε παρατήρηση πάλι. Να πω ότι είναι μια σημαντική έκθεση αυτή η έκθεση. Τα δέματα και οι ταχυδρομικές υπηρεσίε είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μας απασχολεί συχνά, αλλά θα έπρεπε γιατί είναι σημαντικό θέμα επιμελητίας ε, και συνδεδεμένης Ευρώπης. Λοιπόν, η έκθεσή μου έγινε επί τη βάση του ότι ήταν καλή η πρόταση της Κομισιόν, αλλά ήθελε περισσότερη δουλειά και νομίζω ότι και άλλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Το βασικό πρόβλημα εδώ φάνηκε από το ότι πολλοί άνθρωποι, όταν η Κομισιόν εξέτασε την Κομισιόν, είπαν ότι ήθελαν να παραγγείλουν πράγματα ε, στο διαδίκτυο από την Ευρώπη, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κατάσταση των τιμών και την ποιότητα της υπηρεσίας. Είναι λοιπόν ένα θέμα και μεταφορών και καταναλωτών. Και εγώ θεωρώ ότι άρα έπρεπε να δούμε αυτή την πτυχή και τον κλάδο στο σύνολό του. Γιατί αν εστιάσουμε μόνο στους ε, παρόχους ε, καθολικής υπηρεσίας, ε, που βεβαίως με αυτούς ασχολείται κυρίως η οδηγία ταχυδρομικών υπηρεσιών, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις περισσότερες χώρες, έχουν α, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας μικρό τμήμα της αγοράς δεμάτων και μιλάμε για μια αγορά η οποία δεν ρυθμίζεται πάρα πολύ. Αν το συγκρίνουμε με άλλα πράγματα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ακόμα και δικαιοσύνη, όπου η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν έχουμε πολλέ ε, πληροφορίε και τα δέματα ήταν προτεραιότητα της ενιαία αγοράς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν γιατί είχαμε πραγματικά εντατικές συζητήσεις με οργανώσεις ε, του κλάδου, καταναλωτές, συνδικάτα. Ξέρω πως ο κύριος Σλίτσκα, ο συνάδελφός, είχε πολύ καλές συναντήσεις και πολλοί κόσμος είχε συναντήσει με πολλούς ανθρώπους πολύ θετικό. Η ΟΚΕ επίσης το εξέτασε, πολύ σημαντικό. Είναι κρίμα το ότι δεν έκανε μια έκθεση η Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά δεν το έκαναν τελικά. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να έχουμε μια εθνική και περιφερειακή προσέγγιση, κάτι το οποίο κάνουν οι προτάσεις μου. Όσον αφορά λοιπόν την, την έκθεση της Κομισιόν, επί της αρχής ε, κοιτάει ολόκληρη την αγορά, αλλιώς δεν θα ήταν δίκαιο και δεν θα μιλούσαμε για ίσους όρους ανταγωνισμού. Οπότε, για τις βασικές διατάξεις πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχουν ε, και υποχρεώσεις ε, παροχής ε, καθολικής υπηρεσίας και το άρθρο 26 ξεκαθαρίζει ότι αν κάποιος παρέχει την δημόσια υπηρεσία πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι εταιρείε αυτέ ε, να κάνουν τη δουλειά του που την κάνουν προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν ε, αποφάσισα να διαγράψω το άρθρο 6 γιατί δεν ήταν δίκαιο. Δημιουργούσε μια κατάσταση όπου οι πάροχοι πακέτων όπου οι πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας είχαν μικρό μέρος της αγοράς ε, και βεβαίως το να ασχοληθούμε μόνο με αυτούς δεν ήταν λογικό. Ξέρω τώρα πως η Επιτροπή ΙΜΚΟ το βλέπει κάπως διαφορετικά και σκοπεύει να το περιορίσει μόνο στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά όσο περισσότερο μιλούσαμε με, τον, με τους ανθρώπους, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγαμε. Τώρα για τις άλλες διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε σωστά τους στόχους και η Κομισιόν είχε κάνει μια καλή αρχή, αλλά στα άρθρα. Πρέπει να εστιάσουμε στους καταναλωτές, όπως είπαν και άλλοι και βεβαίως να έχουμε και αποτελεσματικές ε, και προσιτές υπηρεσίες. Και η έκθεσή μου στο άρθρο 1 έχει έναν πιο ξεκάθαρο ορισμό για να υπάρχει καλύτερη χρήση της προσβασιμότητας για αποτελεσματική και προσιτή διασυνοριακή υπηρεσία δεμάτων. Και βεβαίως εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για το διασυνοριακό τμήμα. Και βεβαίω εντάξει, μπορεί τα υπόλοιπα να σα φαίνονται κάπως εκτεταμένα, να έχετε κατά νου ότι είχαμε αρκετές παρεμβάσεις εδώ και κάποιες δάνε ακόμη περισσότερες, όπως πλαφών στι τιμέ ή ενιαία ευρωπαϊκή τιμή. Εμείς θεωρούμε λοιπόν πως ε, Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει αργότερα εάν ε, δεν ε, λειτουργήσει το σύστημα. Και έχοντας κατά νου πως η Κομισιόν εν τη σοφία της αποφάσισε και έχοντας εξετάσει όλα τα ζητήματα πως η σχετική οδηγία για την ε, ώρα δεν θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον, αλλά όχι τώρα. Οπότε, στο άρθρο 3, νομίζω πως η Κομισιόν έχει δίκιο όταν ζητάει καλύτερε πληροφορίε και από τις εθνικές Αποπτικές αρχές και αντιλαμβάνομαι πως είναι πολύ εκτεταμένε οι προτάσει μου, αλλά νομίζω πως τι ε, συζητήσεις ε, μπορούμε να καταλάξουμε σε μια σωστή λύση. Λοιπόν, τώρα για τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός και να το γνωρίζουμε όπως ξέρουμε ακριβώς τα δεδομένα για τον τζίρο και άλλα δεδομένα. Και αυτό βεβαίως το είπαμε και στο Συμβουλίο. Και αφορά και τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι πλήρους απασχόλησης, γιατί γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η αγορά αυτή στην πράξη. Επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε δεδομένα για τις διασυνοριακές τιμές ε, και τα τερματικά τέλη και ξέρω πως είναι ένα επίμαχο ζήτημα αλλά είναι μέρος της συνολικής εικόνας και αν οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές ε, είναι και τμήμα του πώς θα αξιολογήσουμε αν έχουμε προβλήματα ανταγωνισμού, προβλήματα με το επίπεδο των τιμών και το αν είναι προσιτές. Αυτή ήταν η άποψη οι δικοί μου, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν συμφωνούν όλοι, αλλά έχουμε έρθει εδώ για να ακούσουμε. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση της προσιτότητας των τιμών, αυτό το δεν λέμε ότι όλοι οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν καθολική υπηρεσία. Αυτό το οποίο κοιτάμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ακριβώ να κοιτάνε τα δικαιώματα μεμονωμένων χρηστών, ε, μικρών επιχειρήσεων, ε, χρηστών οι οποίοι δεν ε, στέλνουν μεγάλες αποστολές όσο είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, ανάπηρους κτλ. Και δεν θεωρώ ότι οι ρυθμιστικές αρχές το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή όπως θα έπρεπε. Και παραμείως, εάν δεν περιλάβουμε το τι κάνουν όλοι οι παροχοί σε μια συγκεκριμένη περιοχή και επιτρέψουμε στις ρυθμιστικές αρχές να δουν την συνολική εικόνα, δεν θα λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Και εδώ πέρα δεν μιλάμε για ρυθμίση τιμών. Δεν θα ερχόμαστε στο τέλος κάθε έτους για να θα λέμε θα ρυθμίσουμε τις τιμές αυτών των εταιριών. Μιλάμε για μια ετήσια έκθεση, όπως κάνει ε, η Κομισιόν π.χ. ένα πίνακα βαθμολογία για την δικαιοσύνη. Ε, στόχο δεν έχουμε λοιπόν να κατανομάσουμε κάποιον, είναι να έχουμε μια αξιολόγηση η οποία θα προσθέτει ε, στο τι συμβαίνει στην πράξη και θα επιτρέψει στον κόσμο να μπορεί να παραγγείλει δέματα από το εξωτερικό. Και τέλος, εγώ νομίζω ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό και το αναγνωρίζει αυτό η Κομισιόν ότι το θέμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών δεν αφορά μόνο την τιμή αλλά και τις παραδόσεις κτλ. Ε, και τις ζημιές, απώλειες αγαθών, επιστροφές κτλ. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν πως ε, στην οδηγία περί προστασίας των καταναλωτών υπάρχει υψηλό επίπεδο αλλά δεν επαρκεί για τον συγκεκριμένο κλάδο και δεν λειτουργεί στην πράξη. Και μας λένε οι καταναλωτές ότι πολλές από τις εταιρείε ηλεκτρονικού εμπορίου δεν παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Και δεν ενδιαφέρονται και για απαιτήσει τυποποίησης. Οπότε δεν είναι τίποτα το ριζοσπαστικό αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα. Λέμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να παρέχονται ε, επιπροσθέτως από την προστασία των καταναλωτών, αλλά να προωθήσουμε και την τυποποίηση και για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί εδώ και 10 χρόνια έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και η Κομισιόν λέει ναι, υπάρχουν διάφορες βέλτιστες πρακτικές, αλλά χρειάζεται μία όφηση. Μπορούσα να πω και άλλα για να εξηγήσω την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, οπωσδήποτε είμαι στην διάθεση των συναδέλφων να συζητήσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι μπορούμε να διαγραφεί τελείως το άρθρο 6, αλλά πέρα από αυτό Νομίζω πως η Κομισιόν έχει κάνει καλή δουλειά. Μπορούμε να συνεργαστούμε εδώ και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντερσον για την σφαιρική αυτή παρουσίαση της έκθεσής σας. Που σίγουρα ε, είναι σημαντική και πρέπει να δοθώ συγκεκριμένε απαντήσει, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα του καταναλωτέ, όπω είπατε και εσείς. Θα ακούσουμε πρώτον λοιπόν τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Φέρμπερ. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, γιατί τα καταφέρνω κάπως καλύτερα από ότι στα ε, γαλλικά για αυτό το πολύ σημαντικό και δύσκολο θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι με εξέπληξε όταν διάβασα το σχέδιο έκθεσης σε ό,τι αφορά αυτή την ανακοίνωση της ε, ε, οδηγίας από την Κομισιόν για ε, τις τραχυδρομικές υπηρεσίες, φανταζόμουν ότι η συγγήτρια θα ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική γραμμή σε σχέση με την ομάδα από την οποία προέρχεται και απογοητεύομαι διότι είχαμε συμφωνήσει μια γραμμή που τώρα την εγκαταλείπει η συγγήτρια. Γιατί, διότι πρώτον το θέμα είναι διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Δηλαδή δεν μιλάμε για, τις, για μια οδηγία σε ό,τι αφορά τις ε, ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες. Δεν προβλέπει κάτι κομισιό συγκεκριμένα για τις ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες, για την, για την αλληλογραφία. Επίσης δεν θέλει να αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά την καθολική υπηρεσία, τις παρόχους καθολικής υπηρεσίας. Και διερωτώ με τώρα όταν διαβάζω αυτό το σχέδιο έκθεσης, γιατί τώρα στον τομέα των δεμάτων που μέχρι τώρα και από το 92 και σε όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ετών έχουμε πει ότι λειτουργεί και δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ο οποίος λειτουργεί γιατί τώρα ε, το ε, αλλάζουμε την, τη θέση μας αυτή. Να μειώσουμε δηλαδή τον ανταγωνισμό. Εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός. Τι να πω. Ε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Έπειτα έχουμε το ερώτημα πού είναι το πρόβλημα και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να εστιάσουμε εκεί. Το πρόβλημα είναι οι τιμές για τα διασυνοριακά πακέτα, για τη διασυνορική παράδοση δεμάτων. Τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσει, ε, Δεν θέλουμε να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό. Ας δούμε την αλυσίδα παραγωγής και αν τη δούμε βλέπουμε ότι το σύστημα μπορεί να πει κανείς ότι ναι με ικανοποιεί, αμοιβέ. Ε, ε, δεν έχουμε πρόβλημα τις καταληκτικές ε, τιμές χρεώσεις κτλ. Ή δεν μου αρέσει και θέλουμε να το αλλάξουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. μπορούμε να αλλάξουμε την παγκόσμια ταχυδρομική σύμβαση. Αν θέλουμε να βάλουμε εδώ και τα σχετικά με την παροχή καθολικών υπηρεσιών για να λύσουμε το πρόβλημα, τι να σας πω, καλή επιτυχία, κυρία Άντερσον. Να σας ε, παραπέψω στις οργανώσεις και τους ενδιαφερομένους, διότι πραγματικά νομίζω ότι οδεύουμε προς καταστροφή ενώ πρέπει να απαντήσουμε άλλα ερωτήματα. Στη δική μου έκθεση ε, είχαμε αφήσει εκτός το ποιος πληρώνει για τις ε, καθολικές πίσεις και τα όλα αυτά τα αφήσαμε εκτός. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει το θέμα των εποπτικών αρχών. που λέτε ότι θα διαφωτίσουν τα περί των, το ελέγχου των τιμών και θα ασχοληθούν με αυτές τις πτυχές. Εμείς αυτό που έχουμε νομίζω είναι το πώς εφαρμόστε και αν εκτελείται το υφιστάμενο δίκαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. αυτοί που έχουν τον έλεγχο ουσιαστικά των τιμών έχουν και τις, ε, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι να ενισχύετε αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο και του άλλους καταστρέφετε. Και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να παρέμβουμε στην αγορά η οποία λειτουργούσε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα, υπήρχε ανταγωνισμός. Δεν το καταλαβαίνω και το ίδιο ισχύει και για την ε, κερδοφορία και την αποδοτικότητα. Εγώ το μόνο που μπορώ να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας ε, που προβλέπει να διευθετήσει το ζήτημα και να μην δημιουργήσουμε μια αγορά που δεν θα δημιουργεί. και κάποια άλλα θεωρητικά ζητήματα. Δεν έχουμε πρόβλημα με το business to business, αλλά διασυνοριακά στο private to private λειτουργεί. Πάμε στο εξωτερικό να σπουδάσουμε, μας στέλνει σπιτικό φαγητό για γιαγιά μας ή γλυκά για να μην πεινάσουμε. Αυτό τι είναι, private to private και διασυνοριακό. Και εδώ το μοντέλο αυτό δεν λειτουργεί. Είναι ε, εκτός και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων το είχα πει. Πού είναι τα δικαιώματά μας καταναλωτή. Με την πρότασή σας, αντί να τα ενισχύετε αυτά τα δικαιώματα, τα αποδυναμώνετε. Αποδυναμώνετε και εμένα τον καταναλωτή και τους παραδοσιακούς παρόχους υπηρεσιών. Και νομίζω ότι πραγματικά δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Θα περιμένω και τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις Είχα κατά νου να καταθέσω κάποιες τροπολογίες, τώρα θα καταθέσω περισσότερες. Πραγματικά πρέπει να πω στην εισηγήτρια ότι με αυτές τις προτάσεις που έχει καταθέσει, αντί να δημιουργεί κάτι, καταστρέφει κάτι. Δημιουργεί, καταστρέφει τις δομές που υπάρχουν. Και δεν είμαστε δετεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Πηγαίνετε με, ε, σε εντελώς λάθος κατεύθυνση με τις προτάσεις και ελπίζω ε, να είναι της ίδιας άποψης ε, και η Επιτροπή. Είναι ρηψοκίνδυνο και παρακινδυνευμένο, γιατί πραγματικά θα ε, προξενήσουμε μεγάλη ζημιά, θα υπάρχουν ολιγοπόλια, να πω μονοπόλια στα κράτη-μέλη, θα αυξηθούν οι τιμές και πραγματικά έχω αφιβολίες για το τι μπορεί να πετύχει η πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Φέρμπερ. Ο κύριος Λοτόφσκι τώρα έχει το λόγο. Μα λέγει τι φεύγετε όμως. Σας παρακαλώ πολύ ξανακαθίστε. Ναι, ναι, η σειρά σας είναι κύριε Σλοτόφσκι. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεσης. σχέδιο έκθεση, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί λαμβάνει υπόψη του πολλά από τα ζητήματα τα οποία θίξαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης μας συζήτησης. Το σχέδιο έκθεση λοιπόν της κυρίας Σάντερσον ανταποκρίνεται και αναφέρεται στις βασικές προκλήσεις όσον αφορά για παράδειγμα την ενίσχυση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι καλύτερη από το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 6. Μπορώ να καταλάβω την πρόθεση που έχει η εισηγήτρια για τη βελτίωση της κατάστασης των καταναλωτών, να μπορούν να έχουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές. Δεν πρέπει όμως να επικεντρωθούμε μόνο στο κόστος. Το ζήτημα τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώ επίση και η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι ζητήματα εξίσου σημαντικά. Τώρα, η επέκταση του πεδίου εφαρμογή σε όλου του φορεί εκμετάλλευση, όλου του παρόχου τέτοιων υπηρεσιών, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλωσορίσουμε. Αυτό προβλεπόταν στο άρθρο 4. Αν δεν υπάρχει επέκταση του πεδίου εφαρμογή σε όλου του αρμόδιους φορεί. δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικέ υπηρεσίε διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Και αν θέλουμε οι υπηρεσίες αυτές να είναι πιο αποτελεσματικέ, τότε θα πρέπει να έχουμε και συλλογή δεδομένων και από του πιο σημαντικού φορεί, τι σημαντικότερε επιχειρήσει. Η κυρία Άντερσον επίσης έθεσε κάποιες ρεαλιστικές προθεσμίε και τροποποίησε αυτές τις οποίες πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προθεσμίες υποβολής ε, στατιστικών δεδομένων προς τις αρμόδιες αρχές. Το άρθρο 5 επίσης θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο και να το τροποποιήσουμε σε σχέση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα άρθρα 5 και τα άρθρα εκείνα που έχουν να κάνουν ε, με την ε, με τον έλεγχο προσιτότητος των διασυνοριακών τιμολογίων, δεν ξέρω τα όσα προτείνει η συγγήτρια είναι πραγματικά ρεαλιστικά και αν δεν θα προκαλέσουν τελικά μεγαλύτερη αναστάτωση στην αγορά. Προβλέπονται εδώ πέρα κάποια χαμηλότερα κατόφλια όσον αφορά τις εξαιρέσεις υποβολής δεδομένων. Προβλέπονται εδώ πέρα κάποια νέα κατόφλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληρώνει 50 μάλλον συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 50 και πάνω από 50. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε περισσότερο την πρόταση της εισηγήτριας, η οποία προτείνει υποχρεώσεις λιγότερο γραφειοκρατικές και λιγότερο επώδυνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό επίσης να αποφύγουμε οποια, οποιαδήποτε αύξηση του κόστους, καθώς επίσης και του γραφειοκρατικού άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές πληροφορίες απαιτούνται, κυρίως όσον αφορά τις καταλεκτικές χρεώσεις. Αυτές οι πληροφορίες όμως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς εμπιστευτικότητας απόρριτου για τις πληροφορίες αυτές. Συνοψίζοντας, χαιρετίζω τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η συγγήτρια, θα έλεγα ότι το έγγραφο αυτό που έχουμε πλέον είναι λιγότερο γραφειοκρατικό σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μένει περισσότερο στα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα αποβάλουμε όμως και κάποιες τροπολογίες. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Στοτόφσκι. Ο κύριος Στέλιτς κάτω έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο, από δύο εναλλακτικέ πλευρέ ουσιαστικά μπορούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό. Είτε να αφαιρθώ σε όλα τα σχετικά ζητήματα που θέλω να θίξω, αλλά δεν πρόκειται πότε να μου δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο, γιατί θα μπορούσα να μιλάω για πολλά λεπτά, ή μάλλον καλύτερα να επικεντρωθώ σε κάποια πιο σημαντικά σημεία. Μπορώ να πω ότι έχω ήδη δει ορισμένους συναδέλφους και θα έλεγα περισσότερο εκπροσώπους από διάφορες οργανώσεις, διάφορους εμπλεκομένους θα θέλετε στον κλάδο αυτό, με τους οποίους έχω συνομιλήσει για τις διατάξεις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά από τις επαφές αυτές που είχα, τους είπα ότι θα αξιολογούσα περισσότερο την προτινόμενη αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση και ότι θα έκανα και κάποιες τροπολογίε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμω να σα αναλύσω με κάθε λεπτομέρεια της παρατηρήσει μου. Συμφωνώ με τους προαλήσαντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Άντερσον. Σίγουρα το ζήτημα είναι αρκετά πολύπλοκο όπως και άλλα νομοθετήματα τα οποία συζητάμε εδώ αλλά θα έλεγα ότι τα υπόλοιπα νομοθετήματα θέλετε προκύπτουν πολύ πιο συχνά και είμαστε πιο εξοικειωμένοι με αυτά. Πρώτη φορά ασχολούμαστε με το ζήτημα αυτό, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε τα ενδιαφερόμενα μέρη, Ποτέ δεν είδα τέτοια μεγάλη απόκληση απόψεων. Πρώτη φορά για ένα τέτοιο ζήτημα βλέπω τέτοια διάσταση απόψεων. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα θυμάστε ενδεχομένω ότι όταν κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια τη Επιτροπή μα για το ζήτημα αυτό, σα είχα πει ότι ήμουν αρκετά διστακτικό και ότι δεν θα μπορούσα εύκολα να συμφωνήσω με μια τέτοια νομοθετική πρόταση. Σήμερα θα σας έλεγα ότι όντως χρειαζόμαστε τελικά μία νομοθετική πρόταση, πρέπει να αξιολογήσουμε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όντως βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Ενδεχομένως να μην συμφωνήσω με κάποιους συναδέλφους. Εγώ δεν ήμουν εισηγητή ούτε σκιώδη εισηγητή για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Ενδεχομένω αυτό να είναι και ατού, δεν ξέρω. Πάντω, από τότε που συζητούσαμε τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε μέχρι σήμερα, το όλο περιβάλλον έχει τροποποιηθεί εντελώ. Πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε ένα μια τεράστια ποσότητα δεμάτων τα οποία αποστέλλονται και πρέπει να δούμε επίσης και πόσο ανταγωνιστική είναι η η αγορά. Όλες αυτές τις παραμέτρους δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια. Παρ' όλα αυτά το επιχειρηματικό περιβάλλον τροποποιείται συνεχώς και βλέπουμε ότι πέρα από τους παραδοσιακούς φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων έχουμε και πολλούς νέους παρόχους, πολλά νέα επιχειρηματικά μοντέλα, μοντέλα όπως η Amazon. Αλλά σε 2, 3, 4 χρόνια ακόμα και για αυτούς τους καινοτόμους αν θέλετε παρόχους τέτοιων υπηρεσιών η κατάσταση θα έχει εντελώ τροποποιηθεί. Χωρίς λοιπόν να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένες διατάξεις επί των οποίων όλα τα διαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πληροφοριών, καλύτερη ενημέρωση. Και αναφέρομαι εδώ πέρα όλους ιδιαίτερα στο άρθρο 3. Και θα ήθελα να δω βέβαια και ποια είναι η άποψη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών επ' αυτού. Επίσης, για να σας δείξω πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα, οι συνάδελφοι μίλησαν για τους καταναλωτές. Σε ποιους καταναλωτές όμως αναφερόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναφερόμαστε σε εμά ως ιδιώτες που αγοράζουμε κάτι διαδικτυακά ή αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να αποστέλουν μεταξύ τους δέματα και να κάνουν χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Σίγουρα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική αυτή η αγορά Μα δίνει ορισμένε φορέ η εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτε οι οποίοι έχουν ηγετική θέση στην αγορά. Σε κάποιε περιπτώσει έχουν ένα περιορισμένο περίδιο αγορά όμω, σε άλλε περιπτώσει έχουν ένα ισχυρότερο μερίδιο στην αγορά, αλλά και οι αγορέ μεταξύ του διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, όντω θα πρέπει να εφαρμοστεί η φυστάμενη νομοθεσία, αλλά τίθεται και το ζήτημα τη επεξεργασία αυτή τη πρόταση. Διαφωνώ με διάφορα σημεία με το σχέδιο έκθεσης και διαφωνώ σε ορισμένα σημεία και με τους συναδέλφους. Πάντως θα συνεργαστώ με τους υπόλοιπους συναδέλφους με τρόπο οικοδομητικό και θα υποβάλω τροπολογίες που πιστεύω ότι θα συμβάλλουν τελικά στη δημιουργία μιας αγοράς η οποία θα λειτουργεί ομαλά χωρίς να δημιουργεί εμπόδια αλλά καταρρύπτοντας τα εμπόδια αυτά και τροπολογίες οι οποίες θα προσβλέπουν στη μελλοντική μορφή που θα έχει αγορά σε 4-5 χρόνια. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Τέλητσκα. Δεν μείνει πολύ χρόνο ε, Πρέπει να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν καλό να μην μακρηγορήσετε και πολύ. Κύριε Γκονζάλη, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομη. Σε γενικές γραμμές θέλω να ευχαριστήσω την συγκήτρια. Το σχέδιο έκθεσης θεωρώ ότι να αξιοποιεί τα θετικά σημεία της πρότασης της Κομισιόν και ενσωματώνει και κάποια στοιχεία από τον οποίο δεν έχει νόημα να έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για διασυνορική παράδοση δεμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και να αναγνωρίσω τις προσπάθειες της Γητεριάς που θέλει να δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια στις βασικές έννοιες του κανονισμού. Και επίση ε, γιατί προτείνει συγκεκριμένε και ενδιαφέρουσε βελτιώσει ε, για του τομεί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παράδοσης των δεμάτων και ιδίως για τις υποχρεώσεις ε, πληροφόρησης που πρέπει να υπέχουν. Υπάρχουν σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε βέβαια. Πρώτον, ο βασικός στόχος του κανονισμού, να μην το ξεχνάμε, είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ε, φορέων που δραστηριοποιούνται στην παράδοση θεμάτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Μόνο το 1-10% όπως των ε, τελών ε, και καταληκτικών χρεώσεων παρουσιάζουν πρόβλημα αδιαφάνειας, άρα πρέπει πιστεύω να θεωρήσουμε ότι καλύτερα αντί να έχουμε ένα πίνακα και όλα αυτά που προτείνονται να εστιάζουμε στις ε, προτάσεις, στις ε, περιπτώσεις εκείνες που έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες ανομοιογένειες. Έχουμε τους μεγάλους ε, ιδιωτικούς ε, φορείς που έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο της διεθνούς αγοράς που είναι και πολύ πιο ευέλικτοι, διότι δεν χρειάζεται να διατηρούν ενεργά τα δίκτυα διανομής για να παρέχουν καθολικές υπηρεσίες στην εθνική, στην εθνική επικράτεια. Και αυτό που κάνουν για να, έχουν, να είναι πιο ανταγωνιστικοί συνήθω ε, πιέζουν προς τα κάτω τους μισθού και υποβαθμίζουν τις ε, συνθήκες εργασία. Άρα, θεωρούμε ότι όλες οι υποχρεώσεις ε, για το μελλοντικό κανονισμό θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους μεγάλους και προς που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό και να εφαρμόζεται σωστά η ισχύουσα νομοθεσία. Ίσως κάτι που θα θέλαμε να αναφέρεται περισσότερο είναι η προστασία των καταναλωτών που είναι ιδιαίτερως ευάλωτοι απέναντι στα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη και θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκοντζάλης. Κυρία Γιούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία που έκανε στην έκθεση της αυτή. Βλέπουμε βέβαια και κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, κάποια άλλα βέβαια τα οποία πρέπει να τα επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο. Και εμείς θα θέλαμε να προχωρήσουμε και λίγο πιο πέρα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι κάπως περιοριστική. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται σε ένα μόνο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή θα δούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα εκτιναχθεί πραγματικά το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα έχουμε όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για τέτοιες υπηρεσίες ε, διασυνοριακές αποστολής δεμάτων. Νομίζω ότι και αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και στο εσωτερικό των κρατών μελών και σε διασυνοριακό επίπεδο και να έχουμε πάντα θεμητές πρακτικές, θεμετικές, θεμητές συνθήκες συνταγωνισμού. Ο κανονισμό όμω αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά όχι μόνο για τι επιχειρήσει αλλά και για του ίδιου του πολίτε. Και θα πρέπει να διέπεται από πλήρη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και διαφάνεια. Γιατί ε, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει τελικά να πετύχουμε έναν διτό στόχο, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Και αυτό συνάδει επίσης και με την γενικότερη αναδυόμενη τάση ψηφοποίησης των υπηρεσίων αυτών. Βλέπετε ότι όλα ουσιαστικά περνάνε όλο και περισσότερο από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίσουμε τη διανομή αυτή δεμάτων από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Α μειωθεί ο χρόνο διαμονή, α αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη προστασία για το περιβάλλον. Η έκρηξη αυτή, αν θέλετε, αυτών των υπηρεσιών, η όλο και μεγαλύτερη αύξησή του, α μην το ξεχνάμε ότι πολλέ φορέ έχει επιπτώσει και στο περιβάλλον. Αυτή την περιβαλλοντική πτυχή μην την ξεχνάμε, σα παρακαλώ. Ως προς όλα αυτά θα υποβάλουμε και εμείς τροπολογίες. Αυτά είχα να πω και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ την κυρία Γιούτο. Το λόγο υπόλοιπη συνάδελφοι, ο κύριος Πακ. Μπαχ. Πάρα πολύ σύντομα. Ο Μάρκους Φέρμπερ νομίζω ότι είπε πολλά, ανέφερε πολλές από τις ε, φοβίες που μας διακατέχουν. Δεν μπορώ να πω ε, βέβαια ότι συμφωνώ με αυτό που είπε για τους ε, φοιτητές που παίρνουν από την γιαγιά τους γλυκά ή φαγητά, καλύτερα τους στέλνουν λεφτά. Τέλος πάντων. Äh, Δύο πράγματα θέλω να πω που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Η διαφάνεια των τιμών το ένα και νομίζω ότι εδώ μπορούμε και πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερες προτάσεις θεωρούν ότι είναι επιχειρηματικό απόρριτο αυτό η επιχειρήση και το δεύτερο είναι η ε, ελευθερία επιλογής. Ως καταναλωτής κάποιος ε, πρέπει να συνειδητοποιεί ότι δεν έχει καμία επιλογή, καμία ελευθερία επιλογής, έχει να κάνει με μια επιχείρηση Και τώρα το ποια επιχείρηση θα μεταφέρει το δέμα, αυτό το αποφασίζουν μεταξύ τους ε, αυτοί που έχουν παράψει τη σύμβαση και δεν ξέρει τίποτα ο καταναλωτής. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρει η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο ανταγωνισμός. Σίγουρα θα έχουμε εξέλιξη και τα επόμενα χρόνια στο, στην αγορά αυτή. Πρόταση της Κομισιόν με εξέπληξε λίγο το 2019 δηλαδή, να καταθέσει μια έκθεση αξιολόγησης. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχουμε μέχρι τότε επαρκέ πληροφορίες στη διάθεσή μας. Δεν είναι αυτός όμως ο μόνος λόγος, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ε, δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Όπως και η συγγήτρια, κυρία Άντερσον. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Ρεβόντα Λον να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία, η οποία μας επιτρέπει πραγματικά να αλλάξουμε πρότυπο, να αλλάξουμε μοντέλο, μια άλλη προσέγγιση στο όλο κείμενο, προκειμένου να μην έχουμε κάλυψη μόνο των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, αλλά να καλύπτονται όλοι οι μεταφορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων είναι ήδη μια αγορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δημιουργούν εμπόδιο σε έναν ανταγωνισμό που ήδη υφίσταται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, βλέπουμε ότι σε αυτές επικεντρώνεται κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έχουμε ομίλους όπως η FedEx, η UPS που βρίσκονται σε ηγετική θέση το να ζητούμε από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να δημοσιεύουν εμπιστευτικές και στρατηγικές ε, ε, πληροφορίες όπως οι καταληκτικές χρεώσεις. Ουσιαστικά αυτό ευνοεί τους μεγάλους ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις που ανέφερα. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ήδη υποβάλλονται σε πάρα πολλούς ελέγχους και υποχρεώσεις διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά στην δημοσιοποίηση των τιμολογιών τους. Σαφώς θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά υπό το πρόσχημα της διαφάνειας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προωθούμε και να βνοούμε τελικά τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε ευνοϊκότερη τελικά θέση σε σχέση με τους φορείς παροχής καθολική υπηρεσία. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και οι προαλήσει εξέφρασαν μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και προσέγγιση. Εγώ να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με την έκθεση αυτή, η οποία όντω είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Αν κατάλαβα καλά, καταρχά συμφωνήσαμε για μια καθολική υπηρεσία, έτσι δεν είναι. Αυτό όμως ε, δεν αποτελεί δώρο τελικά, ουσιαστικά είναι μία υποχρέωση να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ε, λειτουργία των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Και δεχομένως αυτό να μην ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό από οικονομικής πλευράς. Τώρα ερχόμαστε και μιλάμε για μια δεύτερη αγορά, η οποία παρουσιάζει εντονότατη αύξηση χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μια αγορά η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολύ σημαντικά κέρδη μπορούμε να δούμε τα πράγματα από δύο οπτικές γωνίες. Αφενός μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθότι έχουν καταβάλει τέλη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, ή από την άλλη θα πρέπει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, γιατί και αυτός δεν βρίσκεται στην καλύτερη, ε, καλύτερη δυνατή θέση. Και λέμε ότι η αγορά από μόνη της, οι συνθήκες συνταγωνισμού θα λειτουργήσουν υπέρ του καρναλωτή. Τα πράγματα όμως φαίνονται να είναι κάπως αντιφατικά αυτή τη στιγμή. Είδαμε ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι ήδη διστάζουν ως προς τις διατάξεις της, του προτινόμενου αυτού κανονισμού. Ακούσαμε επίσης και την ιδιαίτερα απόλυτη άποψη της κυρίας Μπονφουά, η οποία είπε ότι κατά προτεραιότητα θα πρέπει να προστατεύσουμε τους κρατικούς φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, ακριβώς επειδή παρέχουν μια δημόσια τέτοια καθολική υπηρεσία, δεν ξέρω όμως αν θα πρέπει όντως να λειτουργήσει πλήρως ε, το καθεστώς ανταγωνισμού για να βελτιωθούν και οι συνθήκες για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να γνωρίζω τελικά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο από το ένα ζήτημα στο άλλο να περνάμε δηλαδή από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που θεωρούσαμε ότι είχαμε διευθετήσει και επιτυχώς μάλιστα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει διαφορετικές διαστάσεις, μόλον ότι υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στα δύο. Πραγματικά με μπερδεύει ιδιαίτερα η συζήτηση αυτή. Μα θα προσπαθήσουμε να σας διαφωτίσουμε κύριε Ρικέ, μην ανησυχείτε. Η κυρία Ντεμόντε τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια την κυρία Άντερσον για την εξαιρετική της εργασία και γιατί ε, αφαίρεσε αυτή τη στιγμή την ειδική μνήμα που λεγόταν στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, λέγοντας πολύ σωστά ότι θα πρέπει να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την αγορά. Νομίζω επίσης ότι κάθε φορά που μιλάμε για μια τέτοια αγορά που παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να ισχύει κατά τρόπο αναλογικό και να μην δημιουργεί στρεβλώσεις όσον αφορά την παρέμβαση των διαφορετικών φορέων. Επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άκθος και να καταφέρουμε να έχουμε και την απαραίτητη ποσότητα δεδομένων, η οποία θα μα επιτρέπει να κάνουμε μελέτε, χωρί όμω να επιβαρύνουμε επιχειρήσει και καταναλωτέ. Για το άρθρο 5 θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα πρέπει οι εθνικέ αρχέ να είναι αυτέ που θα αποφασίζουν αν θα πρέπει να κάνουν δοκιμέ ε, ε, προσιτότητα των τιμών. Έπειτα, όσον αφορά το άρθρο 6, νομίζω ότι ε, η υφιστάμενη διάταξη προβλέπεται για τον ανταγωνισμό φτάνει. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να γίνει κάποια αλλαγή. Ο κύριο Βάντεν Κάμπ και μετά η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Βάντεν Κάμπ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο έμαθα ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Του μέγιστου. Και αν δούμε τώρα τα όσα λέει η κυρία Άντερσον, ε, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στο θέμα αυτό και φαίνεται ότι το βέλτιστο είναι ο εχθρός του μέγιστου. Και βεβαίω, ποια είναι η διαφορά, όπως είπε και ο Μάρκους Φέρμπερ, μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και των παρόχων της Καθολικής Υπηρεσίας εξέθεσε τα καθήκοντα και τα δύο, και τον δύο. Και βλέποντας τώρα τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5, τότε αυτή η διαφορά πλέον δεν υπάρχει. Και θα πρέπει οι συμμετέχοντες στην αγορά να δώσουν διάφορες λεπτομέρειες για τις ε, τιμές σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και αναρωτιέμαι πραγματικά αν όλα αυτά πρέπει να μπουν σε αυτόν το, σε αυτό το νομοθέτημα. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια διάκριση. Τέλος, είδα πως η κυρία Άντρεσον υπέβαλε μια τροπολογία, την υπαριθμών 61, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ φτωχών, αναπήρων και ανθρώπων σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό είναι το βέλτιστο. Τώρα, πώς μπορούμε να ζητήσουμε από την υπηρεσία δεμάτων να εξακριβώσει το εισόδημα κάποιου πριν τον χρεώσει. Δηλαδή, η βοήθεια στους στοχούς ανθρώπους θα δίνεται κεντρικά από το κράτος στην περιφέρεια, αλλά δεν, έχει, δεν είναι δουλειά του ανθρώπου ο οποίος παρέχει την υπηρεσία δεμάτων. Έτσι, είστε σε λάθος δρόμο, νομίζω. Συνοψίζοντας, λοιπόν, να υπάρξει διάκριση μεταξύ της αγοράς και του παρόχου της καθολικής υπηρεσίας. Ναι, τιμές του καταναλωτή να τις δώσουν βεβαίως, αλλά το ποια είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ Ολλανδικού και Γερμανικού ταχυδρομείου, αυτά είναι εμπορικά. Μυστικά δεν έχουμε καμία δουλειά να τα ξέρουμε και όπως σας είπα έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τροπολογία 61. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο που είπαμε σε σχέση με τον κανονισμό ήταν ένα όχι, να τον απορρίψουμε, διότι δεν καταλαβαίνω σε αυτόν τον ανοιχτό τομέα ε, πώς θα λυθούν αυτά που λέει η Κομισιόν, ενώ ουσιαστικά ε, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι κάποια έλλειψη διαφάνειας στις παραδόσεις. Ε, αν στείλουμε ένα δέμα από την Ισπανία στη Γαλλία, θα πληρώσουμε άλλη τιμή από αν το στείλουμε από τη Γαλλία στην Ισπανία. Πάντως η αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχει ανταγωνισμός και Αρχικά δεν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα με την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Καλή είναι η εκθέση της κυρίας Άντερσον. Λαμβάνει υπόψη ε, όλους τους ε, φορείς, αλλά πρέπει να εστιάσει ε, σε όλους εξίσου και όχι στους βασικούς. Και στο 4 και 5 μιλάμε για όλους τους φορείς. Και διαγράφει το άθρο 6, γιατί υποχρεούνταν οι εξετατεμένη σε ορισμένα τα οποία δεν υποχρεούνταν οι υπόλοιποι. Βέβαια, εξακολουθεί να μην είναι σαφές το μείγμα αυτή η σχέση μεταξύ ταχυδρομικών αποστολών και δεμάτων. Το πρώτο έχει ρυθμιστεί, υπάρχει πλαίσιο. Ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση δεμάτων είναι ένας άλλος τομέας, με άλλες ιδιαιτερότητες. Και σε ό,τι αφορά την... τις ομάδες ε, και τις ε, κοινότητες που λαμβάνονται υπόψη, νομίζω ότι με την ε, ταχυδρομική οδηγία καλύπτουμε τις επιχειρήσεις Επίσης κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί δεν αναφέρονται οι συμφωνίες μεταξύ κρατών. Δηλαδή τελικά αφήνεται στη δεκατική φύση του κάθε κράτους να κάνει ό,τι θέλει. Εναρμονίζουμε χωρίς να αναρμονίζουμε δηλαδή. Και έπειτα διμερείς αυτές τις συμφωνίες. Που ε, ουσιαστικά ε, προστάτευαν αυτήν την αδιαφάνεια. Βλέπω ότι δεν έχουμε πρόοδο σε αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και κατά τα άλλα πρέπει να πω πως ε, αντιλαμβάνομαι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι την αντίφαση ε, τόσο μεγάλη. Μπορούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς και πρέπει να είμαστε άρα αισιόδοξοι. Θεωρώ πως αναφερθήκαν πάρα πολλά θετικά και σωστά πράγματα. Να επανέλθουμε στις αρχικές σκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ακούγονται εδώ και χρόνια για την απελευθέρωση και τη δημιουργία έστω και τεχνητού ανταγωνισμού ο ανταγωνισμός δεν είναι από μόνος του κακός, αλλά δεν ωφελεί, θεωρώ εγώ, αν αναγκάζει να μπουν ε, μικρές εταιρείες στην αγορά με μεγάλες δυσκολίες ε, και αναγκάζονται να πληρώνουν άσχημα τους υπαλλήλους τους. Δεν μπορεί να είναι αυτό, αυτό το οποίο θέλουμε. Θέλω επίσης να πω ε, για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φέρμπερ στην εισαγωγή γράφει εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων πως οι έρευνες ε, θα δείξουν ότι οι δημόσιες ε, τιμές για, οι τιμές οι οποίες δημοσιοποιούνται ε, συχνά για διεθνείς αποστολές είναι τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω από τις εγχώριες αποστολές δεμάτων. Ποιες είναι οι χώρες και οι Κομισιόν πριν γράψει τέτοια έγγραφα, γιατί δεν πάει σε αυτές τις χώρες ε, να επιβάλλει τα όσα πρέπει ως ε, θεματοφύλακας των συνθήκων. Είναι κάτι το οποίο αναρωτιέμαι συχνά και θέλω να πω παραδείγματος χάρη στο άρθρο 60 είναι νομίζω μια απόδειξη για το πώς η Κομισιόν προσπαθεί τεχνητά με νύχια και με δόντια το άρθρο 6 εδώ πέρα παραδείγματος χάρη να φτιάξει έναν ανταγωνισμό. Μιλάμε για ένα τέρας γραφειοκρατίας ε, που δεν έχουμε ξαναδεί. Μιλάμε για τυποποιημένες προσφορές ε, που θα πρέπει να δηλώνονται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές εντός ενός μηνός ε, κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι γραφειοκρατία, περιττή και δεν έχουν κανένα νόημα να δώσουμε την ευκαιρία στις δουλειές να κάνουν, στις επιχειρήσεις να κάνουν δουλειά τους, αλλά όχι με το ζόρι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο προσπαθήσαμε το τροχαίο υλικό με το ζόρι να το πληρώσει ο δημόσιος τομέας. Όχι να σας πω, δεν είμαι κατά του ανταγωνισμού, αλλά ανταγωνισμός για τον ανταγωνισμό και με το ζόρι, όχι, ε, δεν είναι δυνατόν. Και τέλος. Συμφωνώ με όλους όσον αφορά την διαφάνεια, αλλά δεν μπορεί η διαφάνεια να φτάνει μέχρι του σημείου να λέμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν τους νόμους, που έχουν συλλογικές συμβάσεις, που πληρώνουν τους υπαλλήλους τους, να τιμωρούνται και από πάνω. Δηλαδή να τις αναγκάζουμε να παραδίδουν εμπορικά μυστικά το πώς υπολογίζουν τα τέλη για να δώσουν αυτά τα πράγματα στην Κομισιόν και στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή και σε όλο τον κόσμο τελικά. Νομίζω οι δημοσιοποιημένες τιμές ε, εντάξει, αν έχει πρόσβαση εκεί η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, λογικά κατά υπόλοιπα όμως όλα θεωρώ ότι πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση που μοιάζει με μια ευρωπαϊκή παρακολούθηση των τιμών που δεν έχουμε σε αυτή τη μορφή σε κανέναν άλλο κλάδο. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξο ότι θα βρούμε μια λύση και εγώ θέλω να βοηθήσω σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Στέμακα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Καλημέρα σας. Προσωπείτε την Γενική Διεύθυνση GROW. Ακούσατε τις παρατηρήσεις των αγαπητών συναδέλφων, έχουν εντοπιστεί κάποια προβληματάκια. Για πείτε μας λοιπόν και ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές και καταρχά βέβαια την κυρία Λούση Άντερσον, η οποία έδειξε ιδιαίτερη προσήλωση για το ζήτημα αυτό και έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία στην προετοιμασία τη εκθεσή τη. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και του ευρωβουλευτέ εκείνου οι οποίοι πήραν το λόγο και επέβαλαν παρατηρήσει. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα τεχνικό. Συντοποιούμε επίση ότι είναι αρκετά αμφιλεγόμενο για ορισμένου και δεν μας κάνει εντύπωση ότι δεν συμφωνούν τελικά όλοι οι ευρωβουλευτές, αλλά είπε ο τελευταίος ομιλητής ότι στα πλαίσια ενός επικοδοματικού πνεύματος και συνεργασίας θα καταφέρουμε όλοι να βρούμε μια λύση για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, μόνο ότι καταλαβαίνω ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο έχω στη διάθεσή μου θα καταφέρω να τα θίξω όλα τώρα. Τρει-τέσσερι παρατηρήσει και θα είμαι ιδιαίτερα σύντομο, κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρθει να συμπληρώσει την οδηγία για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Η οδηγία αυτή σχεδιάστηκε μία χρονική περίοδο όπου τελικά η αποστολή επιστολών ήταν αν θέλετε η βασική δραστηριότητα, ενώ τα δέματα ήταν ένα πολύ μικρό μερίδιο τελικά τη όλη δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να είχαμε τροποποιήσει λοιπόν την αρχική αυτή οδηγία, αλλά είπαμε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή και είπαμε ότι χρειάζεται μια επιπλέον συμπληρωματική ε, οδηγία, μάλλον κανονισμός, προκειμένου να καταφέρουμε να συμπληρώσουμε την αρχική οδηγία και να την βελτιώσουμε. Δεύτερον, όσον αφορά την διάσταση προστασίας του καταναλωτή, προφανώς συμφωνούμε με την εισηγήτρια, καθώς επίσης και με άλλους ε, ευρωβουλευτές, ότι ο χρήστης ή ότι ο καταναλωτής βρίσκονται στην καρδιά του όλου αυτού εγχειρήματο. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την εργασία των ε, μικρών ιδίω ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής, καθώς επίσης και να ευνοήσουμε την κατάσταση των ιδιωτών και των ε, ευάλωτων πιο ευαίσθητων ομάδων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Αν για παράδειγμα έχετε λάβει ένα δέμα από έναν ε, έμπορο λιανικής και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα επιστροφής που έχετε, είναι πάρα πολύ ωραίο που θα ήταν πάρα πολύ θετικό μάλλον να υπάρχει μια ενιαία τιμή, ένα ενιαίο τιμολόγιο σταθερό, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για την επιστροφή. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Καταγράφουμε τα όσα είπαν οι ομιλητές για μια επέκταση του πεδίου εφαρμογή και στα δικαιώματα άλλων ομάδων καταναλωτών αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να αποφύγουμε το γραφειοκρατικό άχθος ιδίως για τις επιχειρήσεις. Ετέθη τώρα το ζήτημα αν ε, το σχέδιο αυτό κανονισμού θα πρέπει να αφορά μόνο τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ή όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Ας το δούμε διτός. Ένα μέρος του κανονισμού έχει να κάνει με το σύνολο των φορέων εκμετάλλευσης διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και για όλους αυτούς ισχύει ένα κοινό σύστημα επιτήρησης της αγοράς. Οι μεμονωμένοι φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, θα πρέπει να στείλουν συγκεκριμένε πληροφορίες στις εθνικές αρχές, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό ισχύει για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει προφανώς να γνωρίζουμε πρώτα πώς λειτουργεί η αγορά για να δούμε στη συνέχεια αν λειτουργεί σωστά ή όχι ή αν μπορούν να επέλθουν κάποιες βελτιώσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εισάγει υποχρεώσεις για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Στα άρθρα 4 και 5 που έχουν να κάνουν με τις περαιτέρω πληροφορίες και την προσιτότητα είναι ζητήματα τα οποία βλέπουμε στο άρθρο 12 τις ε, οδηγίες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ισχύουν για τους φορεί παροχή καθολικής υπηρεσίας στα άρθρα αυτά αρκεί βέβαια να υπάγονται στις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και θέλουμε ουσιαστικά τα άρθρα αυτά να τα διευρύνουμε ώστε να ισχύουν και για τους υπόλοιπους φορείς εκμετάλλευσης. Δεν λέμε όμως ότι θα πρέπει και οι ρήτρε προσιτότητα και διαφάνεια να ισχύουν για όλου του φορεί εκμετάλλευση, γιατί ουσιαστικά ήδη καλύπτονται από το προηγούμενο άρθρο το οποίο έθιξα. Στο άρθρο 6 που αναφερόμαστε στην πρόσβαση από τρίτα μέρη, θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό είναι θετικό για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε ότι ένα 90% της διασωνοριακής παράδοσης δεμάτων καλύπτεται τελικά από express couriers και από τις μεγάλες επιχειρήσεις ή από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ευνοήσουμε τις μικρές αυτές επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εφιστάμενα δίκτυα τα οποία ήδη χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας προκειμένου και αυτές οι να μπορούν να παρέχουν συγγνώμη, αυτέ οι επιχειρήσεις να μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο εντελώ δίκαιο και θεμητό. Και ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, και προφανώ είμαι στη διάθεσή σα για να συζητήσω περαιτέρω το ζήτημα αυτό και διμερό. Σα ευχαριστούμε πολύ για τι παρατηρήσει σα. Ένα λεπτό τώρα στην κυρία Άντερσον για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ξέρω ότι υπάρχει και άλλη μια συζήτηση, έχουμε λίγο χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι ακούστηκαν πολλέ ενδιαφέρουσε απόψει. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθώ στην κάθε μία ξεχωριστά. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα συνεδρία στο σχεδόν εισηγητών. Η 16η Μαου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να έρθω μεμονωμένα σε επαφή με τον κάθε ένα που πήρε το λόγο σήμερα και είναι πολύ δύσκολο όντω το ζήτημα αυτό. αφού φάνηκε και από την τεράστια, τεράστια διάσταση απόψεων. Ορισμένα ζητήματα μπορούν να αν δούμε την κατάλληλη ισορροπία που μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα στα άρθρα. Μία λύση θα ήταν να ασχοληθούμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία της εμπιστευτικότητας και της διαφάνειας και να τα μεταφέρουμε σε κάποια άλλα σημεία του κανονισμού, ώστε να πετύχουμε την ευκταία αυτή ισορροπία. Να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε κάτι. Ο κύριος Ρικέ έχει απόλυτο δίκιο. Όντω, είναι πολύ δύσκολο να οριοθετήσουμε το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε, γιατί αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε ένα περιορισμένο αριθμό τιμολογίων που μολονότι μπορεί να είναι διασυνοριακά τελικά αποτελούν τμήμα της καθολικής τελικά υπηρεσίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί και πιστεύω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντερσον. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτά, συνεχίζουμε τις εργασίες μας και περνάμε στο σημείο 6, δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, σχέδιο γνωμοδότησης από τον κύριο Βιμ Βαντεγκάμπ, στον οποίο και δίνω το λόγο. Πρόεδρος, σας παρακαλώ πολύ, εφόσον θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, φύγετε χωρίς να κάνετε ιδιαίτερο θόρυβο. Τώρα το λόγο έχει στο τάκτη γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τα διασυνοριακά πακέτα, το θέμα της Λούση Άντερσον είναι απλό σε σύγκριση με τους μουσουλμικούς κανόνες, το Omnibus που θα μας απασχολήσει τώρα. Αφορά λοιπόν μια αναθεώρηση των γενικών δημοσιονομικών κανόνων που περιέχονται σε 18 κανονισμούς ε, και η Επιτροπή Μεταφορών με άση το άρθρο 54 του κανονισμού έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για κάποια από αυτά τα άρθρα αλλά η Κομισιόν θα πρέπει η Επιτροπή Ήτρα, θα πρέπει να γράψει μια γνωμοδότηση, κάτι το οποίο έκανε εισηγητής ο Γέρζι Μπούζεκ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα του και εισηγητές, αλλά και το προσωπικό της Επιτροπής, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς. Μάρτιν Σούλτς λένε. Και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και άλλη μια συνάντηση συζητήσαμε και εγκρίναμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Μιλάμε λοιπόν για την εισαγωγή κάποιων μηχανισμών blending στο μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη και στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που ελπίζουμε να σημάνουν μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις ε, για τις υποδομές μεταφορών. Υπάρχει μια πολύ σημαντική τροπολογία του συναδελφού Ρικέ που αφορά ακριβώ ε, το θέμα του κινδύνου για τα έργα τα οποία έχουν αυτόν τον χαρακτήρα του blending και στα οποία δεν έχει την κύρια ευθύνη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν ε, μια συμβιβαστική τροπολογία για την τροπολογία του κυρίου ε, Ρικέ και λέμε ότι αν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν πρέπει να ασχοληθούν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει τον κίνδυνο έχει εξολογήσει τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης συζητήσαμε για την σχέση μεταξύ δανείων και επιδοτήσεων. Και εκεί πέρα έχουμε διαφορετικές απόψεις εντό του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ των περισσότερων δανείων, αλλά η κυρία Αγιάλα Σέντερ είναι υπέρ των επιχορηγήσεων, οπότε έγινε και εκεί μια ωραία συζήτηση. Τέλος, ε, ζητώ συγγνώμη. Βεβαίω δεν είναι η Μάρτιν Σούλτ ο συνάδελφο, αλλά Μάρτιν Φούξ. Αυτά. Euh, Ξέρω, το κάνατε τη για να δείτε αν έχουμε αποκοιμηθεί ή είμαστε ακόμη ξύπνοι. Μάλιστα. Προφανές, προφανές. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάμπ για την ε, διάθεσή του να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που εν μέρη βέβαια λαμβάνουν υπόψη ορισμένες από τις δικές μας επιφυλάξεις. Δεν είναι ότι μου αρέσουν ε, οι περισσότερο επιδοτήσει σε σχέση με τα δάνεια, κύριε Βαντεν Κάμπ, αλλά γνωρίζετε ότι η βιομηχανία των μεταφορών ζητά ακριβώς να μην μειώσουμε τον προπολογισμό που έχουμε για τις ενισχύσεις. Γι' αυτό έχουμε και τόσε επιφυλάξεις. Μπορεί η Κομισιόν να έχει λόγο, γιατί δεν θέλει να χάσουμε τα χρήματα του ευρωπαϊκού προπολισμού, αλλά με τη, δι, ιδέα, με, την, τη λύση που προτείνει ουσιαστικά είναι σαν ε, να λέει ότι ε, θα πάμε σε αυτή τη μικρή χρηματοδότηση και ενώ μπορούσαμε να έχουμε κάποια κριτήρια, να επιβάλλουμε κάποια ποσοστά, ποσοστώσεις και στο πλαίσιο του ΣΕΦ, και το χάνουμε αυτό, ε, χάνουμε αυτό το προνόμιο. Επίσης στηρίζουμε τις τροπολογίες για το 80-85% για τα πολιτικά προγράμματα, να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό. Η Κομισιό προτιμά να, να γίνουν όλα άπαξ ε, με μιας, γιατί θεωρείται είναι πιο εύκολη διαχείριση. Όμως εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και τα προγράμματα, τα πιο προσαρμοσμένα, τα ετήσια προγράμματα, για να μπορούμε να περάσουμε και κάποιες από τις δικές μας ε, προτεραιότητες, όπως με τα missing links φέτος. Και βέβαια να βελτιώσουμε και την ε, αποτελεσματικότητα του δικτύου συνολικά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, πέραν του να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντενκάμπ για τη συμβαστική του διάθεση, τη συνενετική του ικανότητα και που ε, μας επέτρεψε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, ο κύριος Ρικέ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω πλήθος βουλευτών ε, να έχει παραμείνει στην αίθουσα και ε, είναι αυτοί που φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται για τα δημοσιονομικά. Και βέβαια άμα μείνουμε από μετρητό μετά καήκαμε, τέλος πάντων. Εξαιρετική έκθεση του κυρίου Βαντεν Κάμπ και εξαιρετικό ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε και την όλη συζήτηση μεταξύ των σκιωδών και του ιδίου. Εμείς θα στηρίξουμε όλες τις συμβαστικέ τροπολογίες και προσωπικά εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία που θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία του ΕΤΠΑ ε, για τις μεταφορές. Να μην αποκλείονται μεταφορές από το κεφάλαιο αυτό από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Το χρειαζόμαστε το Ταμείο. Και έχουμε επενδυτικά μέσα, υπάρχουν ε, οι, τα δάνεια κτλ. Άλλη επιτροπή έλαβε την απόφαση, όχι εμείς, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε για να μπορούν αυτά τα κράτη ε, να εποφελούνται από αυτή τη χρηματοδότηση αυτή. Και για την ΕΤΕΠ, ναι, πρέπει να κάνει τη δουλειά της σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, τι θέλουμε, ε, να καλύπτει τον κίνδυνο, τον, αρχικό κίνδυνο. Ε, είναι λίγο υπερβολικό. Όταν επίσης παριθμούμε τα διάφορα είδη επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων. Νομίζω ότι αποδυναμώνουμε τελικά τις διατάξει, γιατί ό,τι δεν περιλαμβάνει στον κατάλογο μας δημιουργείται εντύπωση ότι δεν υπάρχει καν. Ε, Επομένω, καλό είναι να είμαστε πιο γενικόλογοι. δεν θα στηρίξουμε την τροπολογία 26, γιατί η εξάντε εκ των προτέρων αξιολόγηση αυτών των ε, διατάξεων για το blending είναι κάτι που έχετε σε πλήρη αντίθεση με την ίδια την έννοια του blending αυτής της μικτής, της συνδυαστικής χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να έχουμε εκ των προτέρων αξιολόγηση, είναι Και εφιστώ την προσοχή των συναδέλφων, καλή έκθεση, πολύ καλά ε, καθοδήγησα τις όλες τις συζητήσεις ο εισηγητής μας και θα στηρίξουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Απευθύνουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνω το λόγο στον κύριο Μαγάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω και εγώ κάποια λόγια για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και τις τροπολογίες βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά το ανώτατο όριο του blending. Ένα 10% είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο σημαντικός ο μηχανισμός blending, καθώς επίσης και για το ποσοστό του σεφ που θα μπορούσε να δοθεί στο blending. Εμείς θεωρούμε ότι το 10% είναι ένα λογικό ποσοστό. Μας δίνει μια πρώτη σημαντική χρηματοδότηση προκειμένου να δοκιμάσουμε το σύστημα αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε από το ΣΕΦ και τη χρηματοδότηση και να προσελκύσουμε και επενδύσει. Όσον αφορά την θέσπιση των μελλοντικών συνδυαστικών μηχανισμών χρηματοδότηση, αυτό θα αξιολογηθεί στα πλαίσια τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του ΣΕΦ, υπόκειται σε μία εξάντια αξιολόγηση για να δούμε αν απαιτείται ή όχι και θέλουμε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε εκτελεστικές πράξει αναφερόμενοι στο άρθρο 17 του κανονισμού ΣΕΦ. Επομένως θα έχουμε προγράμματα εργασίας, όπως άλλωστε γίνεται και για οποιαδήποτε χρηματοδοτικό μέσο ή για οποιαδήποτε ε, πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η Επιτροπή ΣΕΦ είναι αυτή η οποία θα αξιολογήσει αν χρειάζεται ένα συνδυαστικό μηχανισμό χρηματοδότησης και εφόσον δοθεί έγκριση από αυτή την Επιτροπή τότε θα ισχύσει, θα τεθεί εν λειτουργία. Επίσης, ετέθη ένα ζήτημα του πόσο φιλοπεριβαλλοντικό είναι το ΣΕΦΕΝ. 80% της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη συνδέεται με φιλοπεριβαλλοντικές οικολογικές μορφές μεταφορών όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η εσωτερική ναυσιπλοεία και ετέθηκε το ζήτημα ορισμένων διατάξεων που επηρεάζουν το ΕΦΣΥ εγώ θα αναφερόμουν όμως στην δεύτερη εκδοχή, αν θέλετε, του ΕΦΣΥ και την απάντηση θα τη βρείτε στον τελευταίο, τον νέο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ένα ακόμα σημαντικό σημείο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά την ανώτατη οροφή που θα μπορούσε να τεθεί για τις μεταφορές στο μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναφερόμαστε όμως σε αυτή τη νομική βάση προκειμένου να προσδιορίσουμε τις ε, συζητήσεις για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα 2,5% του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα δοθεί για τον τομέα των μεταφορών. Και αν πάρετε τώρα τις ε, δραστηριότητες μεταφορών που υποστηρίζονται από τον Ορίστο 2020 και από το ΣΕΦ, φτάνουμε περίπου σε ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Επομένως, το 2,5% που ακούστηκε μας φαίνεται εμάς τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό. Δεν ξέρω αν τώρα θα πρέπει να γίνει εδώ η συζήτηση αυτή. Πάντως είμαστε στη θέση για να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση που έχετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, πώς ακριβώς να το πάρουμε. κάθε περίπτωση δίνω πάλι το λόγο στο συντάκτη γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή και ευχαριστώ τους και ηγητές για τα σχόλια. Είμαστε διατεθειμένοι αύριο το πρωί. Είμαστε έτοιμοι πλήρως να ψηφίσουμε αύριο το πρωί σε 9. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Άρα το ακούσατε, θα ψηφίσουμε αύριο στις 9 η ώρα το πρωί, 9 η ώρα ακριβώς. Συνεχίζουμε τώρα τις κυκλισμένων των θυρών. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα. προκειμένου να σταματήσει η μετάδοση της συνεδρίασης μέσω του διαδικτύου και όσοι δεν